We go. Okay, colleagues, we can resume our business. Everyone can take their seats. σας απόγευμα αρχίζουμε. Σημείο 18 της ημερήσιας διάταξης όπου έχουμε έναν ομιλητή από το Διεθνές Κέντρο Εμπορίου Αράντσα Γκονθάλες, εξτελεστική διευθύντρια του Διεθνούς Κέντρου Εμπορίου. Στους συντονιστές σήμερα το πρωί είπαμε για τη σημασία της οικονομικής ανάπτυξης στις αναπτυσσόμενες χώρες, ιδιαίτερα στην Αφρική και φυσικά οι εμπορικές συμφωνίες ε, συζητούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μερικές ε, οδηγούν σε διχογνωμίες. Επίσης στο πρόγραμμα Aid for Trade έχουμε δυσκολίες, αλλά παρόλα αυτά βλέπουμε ότι οι φτωχότερες χώρες ε, ε, δεν έχουν βιομηχανική βάση για το εμπόριο. Καλό θα ήταν λοιπόν να μας πείτε πώς βλέπετε τις, ε, την εργασία σας και τι τάσεις διαγράφονται. Καλύτερες, υπάρχει θέμα ανασφάλειας, η αστάθεια. Τι μπορεί να κάνει το Διεθνές Κέντρο Εμπορίου. Σας ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ την Επιτροπή ΔΕΒΕ που μου δίνει τη δυνατότητα για να σας πω τι κάνουμε και για να ακούσω και από εσάς πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την εργασία μας. Γνωρίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη είναι μεγαλύτερη συνεισφορή στο Διεθνές Κέντρο Εμπορίου. Είμαστε κάπως άτυπη οργάνωση, γιατί έχουμε και μητέρα και πατέρα που ανήκουν σε δύο διαφορετικούς κόσμους. Το 50% κατά 50% ανήκουμε στα Ηνωμένα Έθνη και χρησιμοποιούμε την εντολή μας για να καταπολεμήσουμε και να εξαλείψουμε τη φτώχεια μέχρι το 2030. Όχι να τη μειώσουμε, αλλά να την εξαλείψουμε, που είναι κάτι το πολύ φιλόδοξο. Ε, κατά 50% ε, ανήκουμε στον ε, ΠΟΕ. Πιστεύουμε δηλαδή ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το εμπόριο ως μέσο οικονομικής ανάπτυξης και χρειαζόμαστε την οικονομική ανάπτυξη αν θέλουμε να εξαλείψουμε τη φτώχεια. Πρόοδο στην εκπαίδευση, στην υγεία, στα ανθρώπινα δικαιώματα και ε, αυτοί οι τομείς θα αντιμετωπιστούν αν έχουμε ισχυρότερες οικονομίες έτσι ώστε οι πολίτες να μπορέσουν να ασκήσουν αυτά τους τα δικαιώματα θεωρητικά. Το 80% των εργασιών μας αφορά το κάτω μέρος της πυραμίδας. Μιλάμε για την υποσαχάρια Αφρική, αναπτυσσόμενες χώρες και χώρες που έχουν βγει από μία σύραξη Μπουρκίνα Φάσο, Φίτζι, Μαδαγασκάρι και ούτω καθεξής ε, Αφγανιστάν κλπ. Πρόκειται για χώρες όπου υπάρχει εμπόλεμη σύραξη και ένταση αλλά και που βρίσκονται στην εμπροστοφυλακή επιπτώσεων κλιματικών αλλαγών. Στο Φίτζι εδώ και τρία χρόνια εργαζόμαστε ε, στεναρά για να γίνει μια διαφοροποίηση των, ε, της βιομηχανίας, αλλά δυστυχώς ένας μεγάλος ε, τυφώνας ακύρωσε την εργασία μας στο Φίτζι. Άρα η οικονομική ανάπτυξη στο κάτω μέρος της πυραμίδας είναι πάρα πολύ δύσκολη, είναι επικίνδυνη, δηλαδή ένα μέρος είναι εφικτό και άλλο όχι, αλλά θα πρέπει να υπάρξει οικονομική ανθεκτικότητα. Επίσης εργαζόμαστε σε χώρες που δεν βρίσκονται στο κάτω μέρος της πυραμίδας, αλλά έχουν πληθυσμούς σχετικούς. Όπου υπάρχει διονγκούμενο πρόβλημα με τους πληθυσμούς που είναι πρόσφυγες τώρα, ενώ μέχρι πριν ήταν μία μέση τάξη, μέση αστική τάξη. Και φυσικά με πολλές ε, γυναίκες, με γυναικείο πληθυσμό, ο οποίος δεν εργάζεται. Τι μπορούμε να κάνουμε για αυτές τις χώρες, είτε πρόκειται για χώρες είτε για πληθυσμούς. Για μας υπάρχουν τρεις βασικοί τομείς. Καταρχήν οι μικροεπιχειρήσεις και οι ΜΜΕ γενικότερα. Κάποτε δεν ήταν θέμα τόσο του σύρμου, τώρα όμως καλύπτουμε το 95% των οικονομικών ζητημάτων και ισχύει ανά τον κόσμο αυτό. Δηλαδή το 95% των επιχειρήσεων είναι ΜΜΕ, μικροεπιχειρήσεις και ΜΜΕ. Μιλάμε για ένα 95% και επιπλέον επιχειρήσεων, 70% απασχόλησης και 50% και λίγο παραπάνω του ΟΑΕΠ. Άρα θα πρέπει να ε, βοηθήσουμε τις ΜΜΕ και τις ε, μικροεπιχειρήσεις για να μπορέσουν να μοχλεύσουν καλύτερα την κατάσταση για την ανάπτυξη, για να μην υπάρχουν αποκλεισμοί και γι' αυτό εργαζόμαστε με τις ΜΜΕ για το σκοπό αυτό. Και ένας τρόπος είναι να βοηθήσουμε τις ΜΜΕ διεθνώς. Όταν συμμετέχουν στο διεθνές εμπόριο είναι πιο ανταγωνιστικές και καταβάλουν καλύτερους μισθούς γιατί είναι πιο παραγωγικές. Υπάρχει ε, δηλαδή ένας ε, φαύλος κύκλος ο οποίος μπορεί να είναι και αποδοτικός στη συγκεκριμένη περίπτωση. Υπάρχει μια κυκλική πορεία δηλαδή. Το να γίνουν πιο ανταγωνιστικές σημαίνει ότι θα τονίσουμε ιδιαίτερα στην υποστήριξή τους έτσι ώστε να συμμετέχουν σε παραγωγικές αλυσίδες και αλυσίδες αξιών. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να μιλάμε για προστιθέμενη αξία μέσα στα πλαίσια της αλυσίδας αξιών είτε κανείς βρίσκεται στο βιομηχανικό τομέα είτε στις υπηρεσίες, δηλαδή τα δύο τρίτα των επιχειρήσεων, είτε στον αγροτικό τομέα, θα πρέπει να προσθέσουμε αξία σε αυτές τις επιχειρήσεις. Γι' αυτό μιλούμε για ε, αυτή την αναβάθμιση αξιών και μεγαλύτερη κάλυψή τους. Τώρα, ως προς τις μικροεπιχειρήσεις και τις ε, ΜΜΕ, θα πρέπει να προωθήσουμε αυτή την ε, ανάπτυξη βιώσιμα, κατά βιώσιμο τρόπο, έτσι ώστε να συμμετάσχουν στο διεθνές εμπόριο κατά βιώσιμο τρόπο, για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στους διεθνού, διεθνείς κανονισμούς, γιατί οι καταναλωτές είναι όλο ένα και πιο απαιτητική και επίσης οι ΜΜΕ θα πρέπει να έχουν καλύτερη συνδεσιμότητα με τις αγορές, δηλαδή πρόσβαση στο, στην καταναλωτική πίστη και στο πιστοληπτικό σύστημα με βάση το σύστημα εξωτερικών επενδύσεων για μεγαλύτερη πιστοληπτική ικανότητα έτσι ώστε να γίνουν επενδύσεις στο χαμηλότερο μέρος της πυραμίδας. Το δεύτερο αφορά την εξύψωση του ρόλου των γυναικών. Είπα ότι οι περισσότεροι φτωχοί είναι στις αγροτικές περιοχές και είναι ιδιαίτερα γυναίκες. Και οι οικονομίες που δεν ενισχύουν το ρόλο των γυναικών είναι λιγότερο παραγωγικές, λιγότερο ανταγωνιστικές, αλλά έχουν και ένα χαμηλότερο ρυθμό μείωσης της ε, φτώχειας, γιατί ξέρουμε ότι το σχέδιο δαπονών των ε, γυναικών είναι διαφορετικό από των ανδρών. Αυτό μας το λένε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Παγκόσμια Τράπεζα. Το 90% των δαπανών των γυναικών αφορούν την οικογένεια, ενώ 40% ε, είναι αντίστοιχες δαπάνες των ανδρών. Αν θέλουμε λοιπόν να εξαλείψουμε την ε, μεγάλη αυτή φτώχεια θα πρέπει να εξυψώσουμε και να ενισχύσουμε τον ρόλο των ε, γυναικών στον τομέα της εκπαίδευσης, υγείας και πολιτικής εκπροσώπησης. Έχει γίνει αυτό εν μέρει, αλλά όχι τόσο στον οικονομικό τομέα. Ως προς το εμπόριο, ο ρόλος των γυναικών είναι μικρότερος από αυτόν των ανδρών και γι' αυτό πλήττονται ιδιαίτερα ως προς το εμπορικό κόστος. Άρα θα πρέπει οι γυναίκες να συμμετέχουν στο διεθνές εμπόριο. Οι διεθνείς συμφωνίες θα πρέπει να γνωρίζουν αυτή τη διάσταση των ε, φύλων. Γι' αυτό υπάρχει μία πρωτοβουλία που φέρει τον τίτλο «She Trades», όπου θα πρέπει να έχουμε ένα εκατομμύριο γυναίκες στην αγορά μέχρι το 2020 και σε 7 τομείς που είναι καθοριστική σημασία στο διεθνές εμπόριο, πρόσβαση στην πιστοληπτική ικανότητα, στα δημόσια έργα, συνδεσιμότητα με τις αγορές και ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα που θα πρέπει να λάβει υπόψη τη διάσταση αυτή των δύο φύλων. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει αυτή η συνδεσιμότητα. Και δυστυχώς οι γυναίκες δεν διαθέτουν και δίκτυα συνδεσιμότητας. Ο τρίτος τομέας δηλαδή ως μετά την ενίσχυση των γυναικών και των ΜΜΕ θα πρέπει να ενισχύσουμε και το κάτω μέρος της πυραμίδας, δηλαδή τους πρόσφυγες. Πρόκειται για έναν ολοένα και διονγκούμενο πληθυσμό, όπου η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να ανταποκριθεί στις ανάγκες τους άμεσα αλλά δεν μπορέσαμε να αντιμετωπίσουμε τις μακροχρόνιες ανάγκες τους ως προς τα οικονομικά δεδομένα. Θα πρέπει λοιπόν οι κοινότητες των προσφύγων να συνδεθούν με την αγορά και να διαθέτουν ένα εισόδημα για να έχουν ή να επανακτήσουν την αξιοπρέπειά τους που χάνουν όταν μετατρέπονται σε πρόσφυγες. Θα πρέπει να σας πω και πού μπορείτε να βοηθήσετε εσείς. Η αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ο μεγαλύτερος συνεισφορέας σήμερα από το δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή, είτε πρόκειται για άμεσα εμπορικές ε, επενδύσεις και συμφωνίες, είτε όχι, εσείς μπορείτε να συνεισφέρετε άμεσα και να αφήσετε το αποτύπωμά σας, γιατί ε, αυτό το κάνετε και σε άλλους τομείς. Δεύτερον, θα πρέπει να υπάρχει συνοχή μεταξύ εμπορικής πολιτικής και αναπτυξιακής να δημιουργούνται ευκαιρίες από τις εμπορικές συμφωνίες οι οποίες να μοχλεύονται κατάλληλα και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να μας δείξει πώς θα συνεισφέρει έτσι ώστε να ανταποκριθεί στους στόχους πώς μπορεί να ανταποκριθεί στους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας. Πιστεύω λοιπόν ότι εσείς είσαστε ο μεγαλύτερος αναπτυξιακός παράγων. Έτσι έχει η κατάσταση ανά τον κόσμο, από τη δική μας θέση. Θα θέλαμε να ακούσουμε τα δικά σας σχόλια και θα προσθέσουμε και εμείς τα δικά μας. Σας ευχαριστώ πολύ γιατί είσαστε ένας μεγάλος εταίρος για το Διεθνές Κέντρο Εμπορίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα εισαγωγικά σχόλια. Εγώ θα ήθελα και να κάνω κάποιες ερωτήσεις. Μήπως μπορείτε να μας εξηγήσετε πιο πρακτικά τι ακριβώς κάνει το Διεθνές Κέντρο Εμπορίου στην πράξη. Γιατί εντάξει λέμε μεγάλα προγράμματα σημαντικά που βοηθούν τις γυναίκες ε, κλπ. Όμως πώς διαλέγετε τις χώρες εταίρου σας, ε, αν συμμετέχετε σε μεγαλύτερα αναπτυξιακά προγράμματα. Ε, για παράδειγμα η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα σύστημα ε, στρατηγικής αναχώρα. Πώς ακριβώς κάνετε την επιλογή αυτή στο πλαίσιο του Διεθνούς Κέντρου Εμπορίου. Είστε το κέντρο εμπορίου που πραγματεύεται ζητήματα διεθνούς εμπορίου, διασυνοριακού εμπορίου ή ασχολείστε γενικώ με διεθνή θέματα γιατί μιλήσατε για τις γυναίκες, μιλήσατε για ε, γυναίκες που διαστηριοποιούνται στο ε, μικρής κλίμακας εμπόριο, ασχολείστε με αυτό ή ασχολείστε με μικρές επιχειρήσεις ε, που εμπορεύονται διασυνοριακά και πώς το κάνετε αυτό, μιλάτε για εμπόριο βορρά και νότου, μία, ένα μείγμα ε, όλων αυτών και πώς ε, ακριβώς, ε, τι έχετε ως γνώμονα στην εργασία σας. Θέλει κανείς να πάρει το λόγο. <clears throat> Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση του έργου σας. Αναφέρετε πολλές βασικές αρχές τις οποίες συμμεριζόμαστε κι εμείς εδώ στην Επιτροπή Ανάπτυξης, δραστηριοποιήστε σε τομείς, σε χώρους, σε περιοχές πριν από συγκρούσεις, μετά από συγκρούσεις, στον τομέα της κλιματικής αλλαγής, αλλά και στο θέμα των προσφύγων. Αυτές οι βασικές αρχές, ότι πρέπει να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα και η εκβιομηχάνηση ο, ο, στόχος για την ε, βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά, της βιωσιμότητας, όλα αυτά είναι, είναι σωστά και τα συμμεριζόμαστε. Αυτό που μου λείπει είναι να μου δώσετε παραδείγματα για το συγκεκριμένο έργο που κάνετε. Να σας πω ένα παράδειγμα. Κάναμε μια διαρευνητική αποστολή στο Λίβανο σε σχέση με τους πρόσφυγες και είδαμε εκεί ότι υπάρχουν σχέδια να βοηθηθούν πρακτικά οι γυναίκες. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν, οι δεξιότητες που αποκτούν μέσα από αυτά τα εκπαιδευτικά προγράμματα οι γυναίκες πρόσφυγες στο Λίβανο, πώς θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν όταν επιστρέψουν στις πατρίδες τους. Εμείς είδαμε λοιπόν συγκεκριμένα παραδείγματα. Το ερώτημα μου προς εσάς είναι, εσείς ε, προσπαθείτε να παρέχετε στις οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στη βάση ε, κατευθυντήρες γραμμές, είχατε χρόνο ε, προκειμένου και τους πόρους τους αναγκαίους προκειμένου να υλοποιήσετε μια τέτοια κατεύθυνση. Ε, να απαντήσετε, λέει η Πρόεδρος, σε αυτές τις ερωτήσεις πρώτα και στη συνέχεια θα ακούσουμε και τους άλλους συναδέλφους. Να ε, σας δώσω συγκεκριμένα παραδείγματα. Να σας περιγράψω δύο είδη έργων, προγραμμάτων. Στη βάση, DADAB, είναι ένας καταβλισμός προσφύγων, ένας χώρος όπου ε, υπάρχουν πρόσφυγες στα, στην Νότια Κένια όπου ε, ζει ένα μεγάλο μέρος ε, μεγάλος πληθυσμός ε, Σομαλών εδώ και 30 χρόνια. Έχουμε δοκιμάσει διάφορα πράγματα. Έχουμε εκπαιδεύσει ανθρώπους, έχουμε δώσει επαγγελματική κατάρτιση σε άντρε και γυναίκες. Διαπιστώσαμε όμως ότι αν αυτή η επαγγελματική κατάρτιση δεν μπορεί να μετουσιωθεί σε εισόδημα, είναι πάρα πολύ απίθανο οι άνθρωποι αυτοί να εγκαταλείψουν το DADAB ή να εγκαταλείψουν έστω ε, τα προγράμματα του ΟΗΕ που του υποστηρίζουν. Τι κάναμε λοιπόν. Πρώτα θέλα, θελήσαμε να κατανοήσουμε τι είδους δεξιότητες υπάρχουν στο ΤΑΝΤΑΠ. Το κάναμε αυτό με, ε, σε συνεργασία με μια μικιο, ε, την ε, νορβηγική που δραστηριοποιείται στο ΤΑΝΤΑΠ και που έχει πολύ μεγάλη εμπειρία εκεί σε αυτόν τον καταβλισμό προσφύγων. Εμείς δεν έχουμε. Παρόλα αυτά όμως ε, εμείς έχουμε εμπειρογνωμοσύνη για το πώς μπορεί κανείς να συνδέσει επαγγελματίες με αγορές. Τι κάναμε λοιπόν, δώσαμε επαγγελματική κατάρτιση σε νέους ανθρώπους, σε άνδρες και γυναίκες, στο DADAB, στον τομέα της πληροφορικής. Και έχουμε πλέον βρει μια ομάδα εταιριών που ενδιαφέρονται να αγοράσουν τις υπηρεσίες που προσφέρουν αυτοί οι άνδρες και αυτές οι γυναίκες που εργάζονται από τον καταβλισμό του Νταντάμπ. Τι κάνουν. Επισημαίνουν φωτογραφίες, αρχιοθετούν ηλεκτρονικά αρχεία και φωτογραφίες, μορφοποιούν έγγραφα ψηφιακά. Προσπαθήσαμε και ξεκινήσαμε ε, από τον ΙΟΙΕ στη Γενέβη να δίνουμε οδηγίες Προ τους νέους αυτούς του ανθρώπους τον Ταντάμπ. Και διαπιστώσαμε ότι το πράγμα λειτουργεί. Πλέον βρισκόμαστε στη δεύτερη φάση όπου στην ουσία έχουμε μετατρέψει όλη αυτή τη διαδικασία σε επάγγελμα. Δεύτερον, δεν μπορούμε προφανώ να βοηθήσουμε μόνο τους Σομαλούς πρόσφυγες που ζουν στην Κένια και να αγνοήσουμε τους κενιάτε του ίδιου. Ε, που είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχουμε αντιμετωπίσει και στον Λίβανο. Άρα, εκεί ε, δουλέψαμε με την Ομοσπονδία ε, Επαγγελματιών Πληροφορικής στην Κένια, ώστε να αναπαράγουμε αυτό το πρόγραμμα το οποίο εφαρμόσαμε στον καταβλισμό Νταντάμπ στο Ναϊρόμπι σε έναν κόμβο πληροφορικής που δημιουργήσαμε εκεί. Τι κάναμε λοιπόν. Οι νέοι άνθρωποι που ζουν στον Νταντάμπ μπορούν πλέον να εγκαταλείψουν τον καταβλισμό αυτό και να επιστρέψουν στη Σομαλία γιατί έχουν πλέον μια, ε, ένα επάγγελμα στα χέρια τους το οποίο μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για να αποκτούν εισόδημα και αυτό και αυτό το θετικό είναι ότι η, δουλειά αυτή είναι και φορητή. Μπορεί κανεί να την κάνει από τον Ταντά, μπορεί να την κάνει και από άλλο μέρο. Δεύτερο παράδειγμα, Καραϊβική. Εκεί υπάρχουν πάρα πολλά μικρά νησιά και πολύ μικρέ και περιορισμένε δυνατότητε προσθήκη αξία. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν πάντοτε κάποιε τέτοιε δυνατότητε. Δουλέψαμε λοιπόν με μια ομάδα εταιριών σε 7 νησιά στον τομέα της καρίδας Πρόγραμμα που χρηματοδοτήθηκε και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρόγραμμα αυτό λοιπόν αφορούσε την μετακίνηση από την εξαγωγή ανεπεξέργαστης καρύδας σε εξαγωγές προϊόντων επεξεργασμένης καρύδας. Τι δηλαδή, νερό καρύδας, λάδι καρύδας, σαπούνι από καρύδα και ο κατάλογος δεν τελειώνει ποτέ. Τι χρειάζεται για να κάνει κανεί αυτό το πράγμα. Πρώτον πρέπει να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα αυτών των μικροπαραγωγών. Πρέπει να μπορούν να παράγουν σύμφωνα με συγκεκριμένα, ε, συγκεκριμένες προδιαγραφές ποιότητας. Που σημαίνει ότι εσεί που είστε ο ενδεχόμενο καταναλωτή αυτών των προϊόντων θέλετε να ξέρετε ότι το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με συγκεκριμένες προδιαγραφέ. Ταυτόχρονα οι μικροπαραγωγοί πρέπει να συνεταιριστούν τους βοηθήσαμε δηλαδή να στήσουν συνεταιρισμούς παραγωγών. Τρίτον, τους φέραμε σε επαφή με επενδυτές και με αγοραστές. Γιατί μεγάλο μέρος της δουλειάς αυτής θα συμπεριλαμβάνει απαραίτητος και επενδυτές προκειμένου να γίνει αυτή η προστίκη αξίας. Αυτές είναι οι αρχές που όπως σας τις περιέγραψα μπορούν να μετουσιωθούν στην πράξη. Περιέγραψα δύο ε, παραδείγματα, αλλά υπάρχει και το κακάο στην Κάνα, στο Εκουαδόρ, μπαχαρικά στην Κασάμπα, στα νησιά Φίτζη, υπάρχει το δέρμα ε, στην Αιθιοπία κτλ. κτλ. Οι βαρχές είναι οι εξής πάντοτε. Δίνουμε σε αυτούς τους παραγωγούς πληροφορίες για την αγορά και την ανταγωνιστικότητα, για να δουν πού μπορούν να διαθέσουν τα προϊόντα τους. Δεύτερον, ενισχύουμε την ανταγωνιστικότητα, συσκευασία, σήμανση κτλ. Τρίτον, υποστηρίζουμε τους θεσμούς τους στην πατρίδα τους, ώστε οι ίδιοι οι θεσμοί των κρατών αυτών να μπορούν να βοηθούν τους παραγωγούς τους ώστε όταν φύγουμε εμείς να μπορούν να συνεχίσουν να αξιοποιούνται οι επενδύσεις που έχουμε κάνει. Τέταρτον, όλο αυτό γίνεται με ολοκληρωμένο και βιώσιμο τρόπο. Εστιάζουμε στους νέους, στις γυναίκες και εστιάζουμε στην βιώσιμη ε, γεωργική πρακτική. Πέμπτον, βοηθούμε τους, ανθρά... ανθρώπους να μειώσουν το κόστος των εμπορικών συναλλαγών με την απλοποίηση των διαδικασιών. Πράγματι, πολλές φορές ε, το εμπόριο ξεκινά σε τοπικό επίπεδο, αλλά στη συνέχεια περνά και σε ένα διασυνοριακό επίπεδο. Και έκτον, αξιοποιούμε τις δυνατότητες ε, του περιφερειακού εμπόριου. Πριν από 30 χρόνια, το εμπόριο, στο εμπόριο το 70% γινόταν μεταξύ των βορείων χωρών. 20% γινόταν μεταξύ βορείων και νοτίων χωρών και 10% γινόταν μεταξύ νοτίων χωρών, χωρών του Νότου. 70-20-10. Σήμερα κινούμαστε σε μια κατεύθυνση όπου το 1 τρίτο των εμπορικών συναλλαγών αφορά τον Βορρά, το 1 τρίτο Βορρά-Νότο και το 1 τρίτο τον Νότο. Άρα οι μεγάλες δυνατότητες σήμερα έγκυνται στο να μπορεί κανείς να συνδέσει τις αγορές του Νότου μεταξύ τους και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και η Βραζιλία, η Κίνα, η Τουρκία είναι μεγάλοι μας εταίροι, σημαντικοί εταίροι του ITC ακριβώς γιατί ε, μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να διασυνδέσουμε τους παραγωγούς και τις χώρες του Νότου. Πώς θα το κάνουμε αυτό ή πώς το κάνουμε ήδη αυτό. Ε, ακολουθούμε μια προσέγγιση και από τα πάνω προς τα κάτω και από τα κάτω προς τα πάνω. Εμείς Είμαστε μια διακυβερνητική οργάνωση και το θετικό είναι ότι το 99% των χωρών ενδιαφέρονται για την αύξηση και τη διεύρυνση των εμπορικών τους δραστηριοτήτων. Γιατί έχουν αναγνωρίσει ότι αυτό βοηθά στην οικονομική ανάπτυξη. Άρα, εμείς εστιάζουμε στις χώρες πολλές φορές εταίροι στην ανάπτυξη μας ζητούν τη βοήθεια γιατί θεωρούν ότι μπορούμε εμείς να υλοποιήσουμε προγράμματα στη βάση. Αυτό συμβαίνει πολύ συχνά με την Ευρωπαϊκή Ένωση για παράδειγμα. Έχουμε εμπειρία 52 ετών, οπότε πολλοί που μας γνωρίζουν έρχονται σε μας και μας ζητούν να συμβάλλουμε στην υλοποίηση των προγραμμάτων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Επίσης, εμείς βοηθούμε όσον αφορά την οργάνωση των εξαγωγών αγωγών. Επίσης, εξετάζουμε το, τις εμπορικές ε, συναλλαγές μεταξύ των χωρών και μας ενδιαφέρει πολύ και η παγκοσμιοποίηση, η διεθνοποίηση των εμπορικών συναλλαγών και των επενδύσεων, γιατί δεν μιλούμε μόνο. Μιλάμε δηλαδή για τέσσερις διατέσεις, διαστάσεις. Εισαγωγές, εξαγωγές και εσωτερικές ε, επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις αν θέλουμε, και αυτό ακριβώς θέλουμε, να μεταρρυθμίσουμε τις χώρες αυτές από τα κάτω προς τα πάνω. Ε, ναι. Μία συμπληρωματική ερώτηση θα ήθελα να κάνω. Με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τι είδους ε, εργασία ε, κάνετε. Είπατε ότι οι οργανώσεις, ε, ότι οι κυβερνήσεις μπορούν να έρθουν και να πούν ε, μπορείτε να μας βοηθήσετε, μπορούν και άλλοι οργανισμοί να το κάνουν αυτό. έρχεστε σε επαφή με το προγραμματισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ποια είναι η σχέση σας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και κάτι άλλο, ε, εκτός από πρόεδρος αυτής της Επιτροπής ε, είμαι και ε, πρόεδρος της ομάδας για το δίκαιο εμπόριο, το Fair Trade στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και υπό την ιδιότητά μου αυτή δεν θέλω να σας κάνω την εξής ερώτηση. Έχετε πολιτικές που σας βοηθούν να υποστηρίξετε αυτές τις οργανώσεις δίκαιου εμπορίου. Μιλήσατε για παράδειγμα για την Καρία και τις ε, μικρές ε, χώρες της Καραϊβικής ε, που είναι παραγωγή των προϊόντων Καρίδας. δεν αφορά όμως ε, μόνο το θέμα του δίκαιου εμπορίου. Για παράδειγμα, στην περίπτωση της μπανάνας καταφέραμε να δημιουργήσουμε, καταφέραμε να δημιουργήσουν μία ε, αγορά ε, γύρω από αυτό το προϊόν και τώρα είναι μεγάλη εξαγωγή μπανάνας σε όλο τον κόσμο. Αυτό είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Πολύ σύντομος θα είμαι. Αναφερθήκατε στην αναπτυξιακή βοήθεια και είπατε ότι ο μεγαλύτερός σας δωρητής είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση Τώρα εμείς ε, προσπαθούμε να επεξεργαστούμε τα διάφορα σενάρια σε σχέση με το Brexit. Ε, κατά τη γνώμη σας πόσο θα επηρεάσει αυτό ε, τον δικό σας οργανισμό και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ποιος θα είναι ο αντίκτυπος του Brexit για την υποστήριξη των προγραμμάτων και των σχεδίων που μας παρουσιάσατε. Ευχαριστώ. Έχουμε εξαιρετικές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, στις διάφορες μεθόδους εργασίας ε, μας ε, σε σχέση με την ανάπτυξη. Έχουμε έναν βασικό συνομιλητή εδώ στις Βρυξέλλες, στην Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, αλλά πολλή αναπτυξιακή δουλειά είναι και αποκεντρωμένη στις διάφορες χώρες. Έχουμε λοιπόν πάρα πολύ καλή σχέση και με τις αντιπροσωπείες στις χώρες και κάθε φορά που πηγαίνουμε επομένως σε μία χώρα, ανεξαρτήτως χρηματοδότησης της ε, συγκεκριμένης ε, προσπάθειας, πάντοτε γνωρίζουμε τους ε, επιτόπου παίκτες και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι βασικός παίκτης όπου και αν πηγαίνουμε σε όλο τον κόσμο. Υπάρχει λοιπόν αυτή η πτυχή και δεν είναι μυστικό ότι αύριο θα, είμαι, ε, θα συναντηθώ με τον Γενικό Διευθυντή ε, της ε, Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης για να μπορέσουμε να καταρτήσουμε μια στρατηγική. Έχουμε επιλέξει δύο-τρει τομεί ε, στου οποίου πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να υποστηρίξει τη δική μα εμπειρογνωμοσύνη και εμεί μπορούμε να υποστηρίξουμε ε, τι προσπάθειε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό το κάνουμε εδώ και πολλά χρόνια με όχι πολύ οργανωμένο τρόπο. Τώρα θέλουμε να οργανωθούμε περισσότερο. Το ξεκινήσαμε ήδη τον περασμένο μήνα με στρατηγικό διάλογο που θα μας δώσει τη δυνατότητα να κάνουμε ένα απολογισμό όλων αυτών των τάσεων που βλέπουμε στην επιτόπου δουλειά μας. Η αηφόρος ανάπτυξη, και λέω για, σε σχέση, απαντάω σε σχέση με την ερώτησή σας για το δίκαιο εμπόριο και πώς αυτό συνάδει με τη δική μας εργασία με την αηφόρο ανάπτυξη. Εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα, το εμπόριο για την αηφόρο ανάπτυξη, ε, που συμπεριλαμβάνει μη κυβερνητικέ οργανώσεις και ιδιωτικές επιχειρήσεις που έχουν ε, προγράμματα για την προώθηση των ε, προϊόντων που προέρχονται από αϊφόρους τρόπους παραγωγής και από αϊφόρες πηγές. Έχουμε όλες αυτές τις προδιαγραφές αϊφορίας. τις έχουμε συμπεριλάβει με ένα, σε ένα συγκεκριμένο κατάλογο. Έχουμε μια ολόκληρη λίστα ε, ε, σωστών ε, προϊόντων και προϊόντων που έχουν παραχθεί με βάση αυτές τις προδιαγραφές που έχουμε θέσει από τα τροπικά δάση μέχρι την έρημο και αυτό το κάνουμε γιατί μπορούν να αποτελέσουν μια βάση εθελοντική για όλους τους παραγωγούς σε όλο τον κόσμο και εμείς βέβαια μπορούμε να ε, συζητήσουμε με βάση αυτές τις προδιαγραφές ε, και ε, με τους τοπικούς παραγωγούς. Έτσι ο συνομιλητής μας δεν είναι μόνο η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης αλλά και Εμπορίου. που αποτελεί ακριβώς μια ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια ε, προώθησης ε, των ε, προδιαγραφών αυτών. Όσον αφορά το Brexit, εμείς και πέρσι και κατά τα επόμενα έτη θα συνεχίσουμε να το κάνουμε εκπονούμε μία έκθεση για την ε, ανάλυση του όγκου, του μεριδίου αγοράς ε, των ε, προϊόντων δίκαιου εμπορίου. Είναι ένας τρόπος που μας βοηθά να καταλάβουμε πού ακριβώς βρισκόμαστε και πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα αποκτήσουν πρόσβαση στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, να του εξηγήσουμε πώς μπορούν να το κάνουν αυτό, όπως το παράδειγμα που είπατε εσείς για την μπανάνα. Αυτό που ακούμε τώρα σε σχέση με το Brexit ε, είναι αστάθεια ε, βραχυπρόθεσμα, γιατί δεν υπάρχει σαφήνεια σε σχέση με το τι θα συμβεί και αυτό δημιουργεί ανησυχίες. Εν μέρη αυτές οι ανησυχίες τις έχει καλύψει το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Υπουργό Εμπορίου πήγε στη Γενέβη την, τον την περασμένη εβδομάδα και είπε ότι ε, οι ε, όροι και προποθέσει που θα ισχύουν για το Ηνωμένο Βασίλειο σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο όταν θα είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα είναι λιγότερο ευνοϊκέ από αυτές που... Ε, ε, υπάρχουν για το Ηνωμένο Βασίλειο στον ε, ΠΟΕ. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό έχει μεγάλη σημασία για ε, τη σχέση των προϊόντων που εισάγονται από το Ηνωμένο Βασίλειο όσο είναι εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, τώρα το κατά πόσο το Ηνωμένο Βασίλειο θα εξακολουθήσει να δαπανά ένα τμήμα του προπολογισμού του, του προπολογισμού του στην αναπτυξιακή βοήθεια, αυτό είναι ένα άλλο θέμα που ετέθηκε. Υπάρχει και ένα ακόμη μεγαλύτερο ερώτημα, ποια είναι η σχέση εμπορίου Ηνωμένου Βασιλείου με ε, την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση όταν ε, θα αποχωρήσει από αυτόν. Αυτό είναι κάτι που δεν έχει λυθεί ακόμη και είναι κάτι το οποίο δημιουργεί ανησυχίε στις ε, υποανάπτυξη χώρες ε, γιατί είναι, υπάρχουν κάποιες ιστορικέ εμπορικές οδοί και ε, ιστορικό εμπόριο και είναι και τμήμα και του, των αξιών τους. Αυτό λοιπόν δημιουργεί ανησυχίες για τους λόγους που εξήγησα. Ευχαριστώ πολύ. Δεν βλέπω κανέναν άλλον να θέλει να θέσει ερωτήματα. Όμω, ο κύριος Καχούνεν από την Γενική Διεύθυνση ΔΕΦΚΟ είναι εδώ. Μήπω θέλετε να προσθέσετε κάτι σε σχέση με ε, τη σχέση αυτή με το Διεθνές ε, Κέντρο Εμπορίου με το ITC. Μήπως θέλετε να μα πείτε περισσότερα πράγματα. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να πάρω το λόγο. Πράγματι, η κοινή εντολή ΠΟΕ και Ηνωμένων Εθνών για το ITC έχει δημιουργήσει μια πολύ καλή φήμη και υποστηρίζει τον ιδιωτικό τομέα και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε αναπτυσσόμενες χώρες, οπότε χαίρομαι πολύ που μπορώ να επιβεβαιώσω ότι έχουμε μια πάρα πολύ καλή σχέση. Έχουμε με το Διεθνές Κέντρο Εμπορίου ένα πολύ καλό ιστορικό συνεργασίας ε, μέσω των διαφόρων προγραμμάτων τοπικών, περιφερειακών αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο ε, και όπως η κυρία Γκονσάλες μας είπε, είμαστε ο μεγάλος ε, δωρητής, εθελοντικά βέβαια, ε, αυτό είχε τα αποτελέσματά του κατά τα τελευταία χρόνια ε, και εξακολουθεί να τα έχει. Τώρα όσο έχουμε να αντιμετωπίσουμε τα, τις προκλήσεις ε, του 2030 και τους υψηλούς στόχους που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από κοινού με το ITC, πρέπει να τονίσω τη συνεργασία μας σε συγκεκριμένους τομείς, στους οποίους αναφέρθηκε και η κυρία Γκονζάλες. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντες αυτοί οι τομείς για παράδειγμα, καλύτερη κατανόηση των αλυσίδων αξιών και των τελικών αγορών, καλύτερος προγραμματισμός και καλύτερος αντίκτυπος, ε, ενδεχομένως πιλωτικά προγράμματα που μπορούν να αποτελέσουν παράδειγμα σύνδεσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με τις αγορές, βελτίωση επίσης ε, του επιχειρηματικού και του ρυθμιστικού ε, περιβάλλοντος στις χώρες αυτές, Βέβαια, σε αυτού του τομεί υπάρχει άμεση σχέση και με το σχέδιο εξωτερικών επενδύσεων. Ε, συμφωνούμε απολύτως ε, με την ε, βαρύτητα που δίνεται στην νεολαία και στην οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών. Με πολύ χαρά λοιπόν θα προσέλθουμε στην αυριανή συνάντηση και θα εξετάσουμε αυτούς τους τομείς ε, στους οποίους μπορούμε να ενισχύσουμε αυτή τη συνεργασία και πραγματικά ε, είναι πολύτιμη για μας ε, η δουλειά του Διεθνούς Κέντρου Εμπορίου. Υπάρχει τίποτα άλλο που θα θέλατε να προσθέσετε, λέει Πρόεδρος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ λοιπόν που ήσασταν μαζί μας σήμερα και που μας είπατε όλα αυτά για τον οργανισμό σας. Ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε σύντομα να ε, δούμε τους ε, καρπούς. Ε, είναι πολύ σημαντικό που σας γνωρίσαμε και όλες και ξέρουμε με ποιον συνομιλούμε. Να ευχαριστήσω λοιπόν την προσκεκλημένη μας, την κυρία Γονσάλες, για την παρουσία της εδώ σήμερα. Περιμένουμε δύο λεπτά. Βλέπω ότι έχει έρθει και άλλος εκπρόσωπος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα οι ομιλητοί να προσέλθουν εδώ. Να έρθετε δίπλα μου. Οι πρώτοι δύο ομιλητές είναι της ε, Επιτροπής. Yeah. Okay, so sorry to ε, ζητώ συγγνώμη από την Ναταλή, από την Oxfam. Έχουμε εδώ χώρο, μπορείτε να έρθετε κι εσείς. Sorry, colleagues, we're waiting for DG DevCo. I thought they were here. We won't let, let DG DevCo arrive because they are the lead. Ε, περιμένουμε και εκπροσώπους από την Γενική Διεύθυνση DevCo. διακόπτουμε για δύο λεπτά μέχρι να έρθει υπεύθυνο.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

Okay, colleagues, thank you for being patient because we wanted to make sure. Λοιπόν, ε, καθυστερήσαμε λιγάκι για να είναι παρόντες και παρούσες όλοι οι ομιλητές. Ε, τώρα θα ασχοληθούμε με το θέμα υπαριθμών 19 ευρω... 14 και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που η κυρία Γέγκερ είναι εδώ μαζί μας. Ο Γιάγκερ, Γιάγκερ, Γιάγκερ, from the Deputy Director General. Ε, λοιπόν, θα μας απασχολήσει το εξωτερικό επενδυτικό σχέδιο και η ε, Κατερίνα Μαλτενόβα από την DG είναι παρούσα που συμμετέχουν σε αυτό το πακέτο μαζί με την κυρία Μαριέτα ε, Γέγκερ μέσα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξωτερικού Επενδυτικού Σχεδίου. Όπως ξέρετε, το Σεπτέμβριο ο πρόεδρος Γιούνκερ ανακοίνωσε το Εξωτερικό Επενδυτικό Σχέδιο για να ασχοληθούμε με το θέμα της μετανάστευσης καθώς και της, ε, των ιδιωτικών επενδύσεων στην Αφρική. Το πακέτο αυτό βρίσκεται ενώπιον της Επιτροπής ΔΕΒΕ. Θα ασχοληθούμε με το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Αϊφόρο Ανάπτυξη όπου γνωρίζετε ότι είμαστε η επικεφαλής ε, επιτροπή και δύο άλλα μέσα που ασχολούνται με το ρόλο της ε, Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Α, μάλιστα, μόλις έφτασε ο εκπρόσωπος από την ΕΤΕ. Και φυσικά Πέρα από την ε, ΕΤΕ, η Επιτροπή Προϋπολογισμών θα γνωμοδοτήσει για τις δύο άλλες εκθέσεις. Εμείς θα ασχοληθούμε με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η Επιτροπή έχει εγγράψει 3,3 δις μέχρι το 2020 και οι συνάδελφοι θα μας πούνε πώς θα χρησιμοποιηθούν αυτοί οι πόροι. Καταρχήν θα ακούσουμε από την Επιτροπή, θα μας παρουσιάσει το επενδυτικό σχέδιο και θα θέλαμε να μας πείτε ποιο είναι το υπόβαθρο της όλης πολιτικής και να μας μιλήσετε και για τεχνικά ζητήματα για να γνωρίζουμε από πού προέρχονται τα χρήματα, ποιες είναι οι προσδοκίες και ούτω καθεξής. Ξέρουμε ότι υπάρχουν ε, μεγάλες δυσκολίες, το έχουμε συζητήσει εδώ και καιρό. Θέματα μετανάστευσης δηλαδή και στη συνέχεια μετά τις ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο κύριος Νικολάη Ντοφγκίλεβιτς εξ ονόματος της ε, ΕΤΕ του Γραφείου των Βρυξελών θα μας απαντήσει σε σχέση με το ρόλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Έχετε μεταβεί στην Αφρική πρόσφατα και ξέρετε ποιος είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Και μετά η Oxfam θα μας πει πώς βλέπουν αυτά τα νέα μέσα και σχέδια από την Oxfam χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση. Θα αρχίσουμε την κυρία Γέγκερ. Μαριέτα Γέγκερ. Να μας πείτε την άποψη της ε, Γενικής Διεύθυνσης ε, ΔΕΒΚΟ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και σας και την Επιτροπή σας γιατί μας καλέσατε για να σας παρουσιάσουμε το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό ε, Σχέδιο Εξωτερικής Πολιτικής. Όπως ξέρετε, τον Ιούνιο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προβλήθηκε ένα επενδυτικό σχέδιο μέσα στα πλαίσια της κατάστασης της Ένωσης που προέβαλε ο πρόεδρος ο κύριος Γιούνκερ. Άρα το εξωτερικό επενδυτικό σχέδιο προβάλλει μια μακροχρόνια προσέγγιση για να προωθήσουμε τις επενδύσεις, διότι οι ευφυείς επενδύσεις και οι βιώσιμες επενδύσεις παίζουν σημαντικό ρόλο στις αναπτυσσόμενες χώρες για τη σταθερότητα και την ε, βελτίωση των καταστάσεων της κατάστασης σε ευάλωτες χώρες. Άρα οι επενδύσεις είναι βασικός τομέας έτσι ώστε να προωθήσουμε την ε, αναπτυξιακή πολιτική και την ε, οικονομική ατζέντα της Μπεμπα καθώς και το ΚΟΠΣ. Θα ήθελα λοιπόν να θυμόσαστε ότι έχουμε ε, να κάνουμε και με ε, επιδοτήσεις οι οποίες όμως δεν μπορούν να ανταποκριθούν στην παρούσα κατάσταση. Θα πρέπει να γίνει καλύτερη χρήση των δημοσίων πόρων. Γι' αυτό το εξωτερικό επενδυτικό σχέδιο θα επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να διαδραματίσει παραδειγματικό ηγετικό ρόλο πέρα από τα κλασικού τύπου σχέδια που είχαμε μέχρι τώρα. Το σχέδιο θα κινητοποιήσει επενδύσεις, θα προωθήσει τεχνική υποστήριξη καθώς και τις οικονομικές και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις είναι ύψης της σημασίας για να προωθήσουμε την μακροχρόνια βιωτική ανάπτυξη. Διαφορετικά, οι επενδύσεις δεν θα έχουν μακρόπνοες επιπτώσεις. Θα έχουμε και έναν τεχνική υφής κανονισμό, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να ε, δελεάσουμε τον ιδιωτικό τομέα και να έχουμε ένα, μία πρόσδεση στις επενδύσεις με χαμηλό κόστος, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις με βάση τη βοήθεια προς ΜΜΕ και ισότητα αντιμετώπισης των δύο φύλων. Θα χρησιμοποιήσουμε και την ΣΟΕΣ ε, με βάση αυτά που είπε και η Πρόεδρος, δηλαδή συνεισφορά 3,3 δις από τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Η Κατερίνα θα σας μιλήσει για τους τρεις πυλώνες και την χρηματοπιστωτική διάρθρωση. Άρα το, το επενδυτικό σχέδιο θα βασιστεί στους τρεις πυλώνες. Καταρχήν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Βιώσιμης Ανάπτυξης που θα ενσωματωθεί σε αυτό το χρηματοπιστωτικό πακέτο και στην ε, πλατφόρμα κοινωνικής ανάπτυξης καθώς και το σύστημα εγγυήσεων που είχαμε από το 2007 μέχρι το 2015. Προσπαθήσαμε και καταφέραμε να καλύψουμε 278 project από το αρχικό ποσό που προβλεπόταν και ήταν της τάξης των 15 δις. Θέλουμε και τη συνδρομή ε, του ιδιωτικού τομέα ε, η Κατερίνα θα σας μιλήσει και για τον τεχνικό πυλώνα στη συνέχεια. Για μας έχει μεγάλη σημασία και ο τρίτος πυλώνας. Δηλαδή το να βελτιώσουμε τον ε, ε, επιχειρηματικό τομέα και φυσικά η αιτιώδη συνάφεια των, τρι, τριών πυλώνων είναι μεγάλη σημασία για μια ολιστική προσέγγιση ως προς τον τρίτο πυλώνα. Έχουμε εδώ μαζί μας και εκπρόσωπο από την Oxfam. Είχαμε μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις που κατέληξαν στις 28 Αυγούστου και με την κοινωνία των πολιτών για να ε, προβάλλουμε έναν διάλογο όχι μόνο σε κυβερνητικό επίπεδο και τον ιδιωτικό τομέα, αλλά και με την κοινωνία των πολιτών. Και είμαστε πεπισμένοι ότι η κοινωνία των πολιτών έχει σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει για την εφαρμογή αυτού του σχεδίου σε κρατικό επίπεδο. Συμβαδίζουμε λοιπόν με τις ανησυχίες της κοινωνίας των πολιτών. Λαμβάνουμε υπόψη τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα ε, ως προς την έγκυο ιδιοκτησία με βάση το εξωτερικό επενδυτικό σχέδιο. Αυτό που μας ενδιαφέρει λοιπόν είναι τα κοινωνικά βιώσιμα σχέδια στο διαρθρωτικό τομέα θα ήθελα καταρχήν να σας πω ότι βασιζόμαστε στα ε, μέσα αλληλεπίδρασης και αλληλενσωμάτωσης, blending facilities, όπως ισχύουν μέχρι τώρα. Σύμφωνα με την πρόταση της Κομισιόν, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορούσε να συμμετάσχει σε μια στρατηγική πλατφόρμα και θα μπορούσατε να συμμετάσχετε και στην αναθεώρηση των στρατηγικών και των στόχων. Είναι ζωτική σημασία να συμμετάσχουν όλοι οι οικονομικοί μηχανισμοί και φορείς. Χαίρομαι που βλέπω τον φίλο Μικαέλ εδώ και αυτό που έχει σημασία είναι να στεφθεί όλο το, το όλο εγχείρημα από επιτυχία. Θα πρέπει δηλαδή να λάβουμε υπόψη και τον ρόλο της ΕΤΕ. Η ΕΤΕ ε, είναι τεχνικός σύμβουλος μέσα στα πλαίσια του Ταμείου Εγγυήσεων και αποτελεί έναν βασικό εταίρο. Θα ήθελα να τονίσω ότι οι δραστηριότητες καθώς και το Ευρωπαϊκό Εξωτερικό Επενδυτικό Σχέδιο ε, λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια επιλεξιμότητας με βάση τις διαπραγματεύσεις δηλαδή που έχουν προωθηθεί και λαμβάνουμε υπόψη τους κανόνες του παραρτήματος 2. Όλα τα ταμεία λοιπόν μπορούν να θεωρηθούν ODA. Τις τελευταίες εβδομάδες το Συμβούλιο έχει ξεκινήσει με την επιλογή των, ε, του σχήματος και όσο γνωρίζω υπάρχει πολύ καλή συνεννόηση για όλα τα σχέδια και τις προτάσεις γιατί υπήρχαν και προωθήθηκαν και τεχνικά σεμινάρια και από το Κοινοβούλιο γιατί πιστεύουμε ότι αυτά τα επεξηγηματικά σχέδια έχουν μεγάλη σημασία έτσι ώστε να αρθούν οι ανησυχίες σας. Σας υποστηρίζουμε λοιπόν και θα σας δώσουμε και τις κατευθυντήριες γραμμές μέσα στα πλαίσια της αποκοινού νομοθέτησης για να εγκρίνουμε αυτό το σχέδιο με τάχιστη διαδικασία. Η Κατερίνα έχει το λόγο. Η Κατερίνα λοιπόν είναι αναπληρώτρια ε, Γενική Διευθύντρια της Γενικής Διεύθυνσης ΝΙΑ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ αξιότιμοι βουλευτές αγαπητή Μαριέτα. Εμείς πιστεύουμε ότι η πρωτοβουλία παρουσίασης του εξωτερικού επενδυτικού σχεδίου έρχεται σε μια πραγματικά πολύ κρίσιμη στιγμή ακριβώς γιατί μας δίνει τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε κάθε ευρώ αναπτυξιακής βοήθειας που δίνει ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός τόσο στην Αφρικανική Ήπειρο αλλά και στις χώρες της γειτονίας. Όπως γνωρίζετε, στην ανακοίνωση του Ιουνίου με την οποία ξεκίνησε αυτή η διαδικασία δημιουργίας του εξωτερικού επενδυτικού σχεδίου δόθηκε μεγάλη έμφαση στο να αντιμετωπιστούν τα ριζικά αίτια της μετανάστευσης κάτι που βρίσκεται και στο επίκεντρο των γενικότερων αναπτυξιακών μας προσπαθειών. Όπως είπε και η Μαριέτα, το εξωτερικό επενδυτικό σχέδιο θεμελιωδώς ε, αποτελεί μια πρωτοβουλία για την ανάπτυξη και αποτελείται από τρεις πυλώνες. Οι τρεις πυλώνες πραγματικά αλληλοδιαπλέκονται και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Ο πρώτος πυλώνας είναι οι επενδύσεις ε, δεύτερος πυλώνας είναι η τεχνική βοήθεια και ο τρίτος πυλώνας είναι ε, το επενδυτικό κλίμα αλλά και το εν γέννη, το γενικότερο κλίμα γιατί, και περιβάλλον. Γιατί ε, χρειάζεται ένα επενδυτικό περιβάλλον το οποίο να μπορεί να αξιοποιήσει τη χρηματοδότηση που δίνεται. Όσον αφορά τον πρώτο πυλώνα, τον απο τον αποκαλέσαμε λοιπόν Ευρωπαϊκό Ταμείο Βιώσιμης Ανάπτυξης, που όπως είπε και η Μαριέτα αποτελείται από δύο στοιχεία. Το πρώτο στοιχείο είναι ότι ε, είναι αυτή, αυτό τον, αυτή η νέα διάσταση των εγγυήσεων που δημιουργήθηκαν ακριβώς για να ξεπεράσουμε ε, την μόχλευση που την ε, ε, επιτυχάνουμε μέσω του δεύτερου πυλώνα και της πλατφόρμας που δημιουργήθηκε ε, για, για, για, τα, για τα καθεστώτα, τα συστήματα, τα αναπτυξιακής βοήθειας για τη Μεσόγειο και την Αφρική. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε με τις εγγύησεις είναι πέραν, πέραν της μόχλευσης να εμπλέξουμε και τον ιδιωτικό τομέα ώστε να κάνει επενδύσεις στην ανάπτυξη για να διασκεδάσουμε και κάποιες από τις ανησυχίες που έχουν ακουστεί. Εδώ δεν μιλούμε για χρήματα που θα δοθούν στον ιδιωτικό τομέα, στον ευρωπαϊκό ιδιωτικό τομέα ως τέτοιο. Πρόκειται για χρήματα για την ανάπτυξη που θα διοχετευθούν μέσω των εταίρων μας, κατά κύριο λόγο βεβαίως μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, αλλά και άλλων αναπτυξιακών ε, τραπεζών και πιστοτικών ε, ιδρυμάτων που θα συνεργαστούν με τον ιδιωτικό τομέα. Ναι, λοιπόν, υπάρχει η δυνατότητα ο ευρωπαϊκός ιδιωτικός ε, τομέας να αξιοποιήσει αυτήν την ε, διαδικασία χρηματοδότησης, αλλά ο πύχης μπαίνει πάρα πολύ ψηλά. Υπάρχουν ισχυρότατες εγγυήσει στον, ε, στο μηχανισμό που έχουμε δημιουργήσει, ώστε να μπορούμε να πούμε με ασφάλεια ότι θα τηρούνται και ε, οι, τα, οι κοινωνικές και περιβαλλοντικές προδιαγραφές ε, όσον αφορά το, την χρηματοδότηση και την αναψυξιακή βοήθεια που θα δίνεται. Από αυτή την άποψη το σεμινάριο που θα γίνει την Παρασκευή και στο οποίο αναφέρθηκε η Μαριέτα θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο για να δοθούν πληροφορίες για το πώς ακριβώς θα λειτουργήσει αυτό το Ταμείο. Γιατί ως προς την νομοθετική ε, πρόταση είναι το μοναδικό στοιχείο στο οποίο θα ε, κληθείτε να συμμετάσχετε στη συζήτηση. Ε, υπάρχει ένα ευρύτατο πλαίσιο. Το νομοθετικό λοιπόν είναι πολύ στενό ε, και το οποίο θα, θα αφορά ακριβώς αυτές τις εγγύησει. γιατί η διαδικασία αλληλεπίδρασης και συγχώνευσης θα αφορά ε, μόλις το, το 20%. Το 80% των προσπαθειών μας αφορά τη συγχώνευση και τον συγκερασμό διαφόρων πρωτοβουλειών και πλατφορμών που θα θα τους δοθεί μια νέα κατεύθυνση προκειμένου να μπορέσουμε να συντονίσουμε καλύτερα το έργο μας με τους εταίρους μας. Και όταν αναφέρομαι σε εταίρους, ενώ την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, άλλες εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες και πιστοτικά ιδρύματα, καθώς και άλλους διεθνείς πιστοτικούς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στη χώρα ε, όπου ε, υλοποιείται κάποιο πρόγραμμα στο πλαίσιο του επενδυτικού εξωτερικού σχεδίου. Με άλλα λόγια, έχουμε ένα σύστημα το οποίο πλέον θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία και που ως προς τους στόχους του θα συμπεριλαμβάνει την αντιμετώπιση των ριζικών αιτίων της μετανάστευσης αλλά ταυτόχρονα θα δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη συνεργασία με τις χώρες από την Αφρική, την ευρύτερη γειτονία και σε όλη αυτή τη διαδικασία θα ε, ε, βρισκόμαστε σε διαρκή και στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κομισιόν, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης αλλά και τους άλλους εταίρους μας. Αυτή λοιπόν είναι δύο, τα δύο στοιχεία, να το πω έτσι, που ε, συναποτελούν αυτό το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη και συγκεκριμένα τον πρώτο πυλώνα. Τώρα, όσον αφορά τον πυλώνα 2, αφορά την τεχνική βοήθεια όπως είπα και όποιος έχει δουλέψει στον τομέα της αναπτυξιακής βοήθειας γνωρίζει ότι αν δεν έχει κανείς την ικανότητα να συνδυάζει δύο πράγματα, δηλαδή και να υποστηρίζει ε, την, ε, την ανάπτυξη έργων και προγραμμάτων σε αδύναμα περιβάλλοντα αλλά ταυτόχρονα να υποστηρίζει και την πολιτική, δηλαδή την χάραξη θετικών πολιτικών που θα δίνουν τη δυνατότητα οι επενδύσεις να αποδίδουν σε δύσκολα περιβάλλοντα είναι αυταπάτη να προσπαθεί κανείς να να νομίζει ότι μπορεί να επιτύχει τους στόχους του αν δεν ακολουθήσει συγκεκριμένους τρόπους, συγκεκριμένες μεθόδους. Γι' αυτό και ο δεύτερος πυλώνας αφορά την τεχνική βοήθεια. Ο τρίτος πυλώνας αφορά το ε, επενδυτικό περιβάλλον, το επενδυτικό κλίμα και το γενικότερο περιβάλλον. Εκεί μιλούμε για ζητήματα αδειοδότησης, διάθεσης προϊόντων στην αγορά, νομοθεσίες κτλ. κτλ. Στο γενικότερο πλαίσιο μιλούμε για τον, τον δημοσιονομικό χώρο, για τις επενδύσεις, για την καταπολέμηση διαφθοράς, για την, ε, τη διαφάνεια. Όλα αυτά δηλαδή που συναποτελούν το περιβάλλον εντός του οποίου μπορούν οι επιχειρήσεις να ανθίσουν και να δραστηριοποιηθούν ε, ε, επιχειρηματικά. Αυτά λοιπόν ε, εντάσσονται όλα στον πυλώνα υπαριθμών 3. Θα τελειώσω λέγοντας δύο λόγια για τη διακυβέρνηση. Εμείς βρισκόμαστε ακόμα στη διαδικασία κατάρτισης ή εν πάση περιπτώσει προσδιορισμού ε, κάποιων τελικών λεπτομεριών όσον αφορά την διακυβέρνηση. Θα υπάρξει σε κάθε περίπτωση μια στρατηγική επιτροπή η οποία θα επιβλέπει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Βιώσιμης Ανάπτυξης δηλαδή και τους τρεις πυλώνες που σας παρουσίασα και ταυτόχρονα ε, η Επιτροπή αυτή θα, έχει, ε, θα διαθέτει και μια γραμματεία, ενώ οι επενδυτικές πλατφόρμες θα ε, διοικούνται από τις επιχειρησιακές επιτροπές. Μιλούμε για δύο γιατί στην ουσία μιλούμε για δύο διαφορετικούς γεωγραφικούς χώρους. Αφενός μιλούμε για την, το επενδυτικό σχέδιο για την Αφρική και το επενδυτικό σχέδιο για τη γειτονία. Αυτά τα δύο σχέδια ε, αφορούν δύο διαφορετικούς γεωγραφικούς χώρους και δύο διαφορετικές ομάδες χωρών. Θα υπάρχει λοιπόν μία γραμματεία, μία καινιαία γραμματεία η οποία θα ενοποιεί το έργο και η Στρατηγική Επιτροπή θα έχει την ευθύνη ελέγχου της συνοχής του όλου συστήματος που δημιουργούμε. Όσον αφορά τη χρηματοδότηση, το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη θα έχει 3,35 δισεκατομμύρια ευρώ στην διάθεσή του, εκ των οποίων η εγγύηση είναι 1,5 δις. 750 εκατομμύρια είναι η συμβολή από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τα οποία συνδυάζονται άλλα 750 εκατομμύρια ε, που θα μοχλευθούν από την ε, οικονομία και ελπίζουμε τα κράτη-μέλη να σταθούν αρρωγοί σε αυτήν την προσπάθεια, γιατί προκειμένου να επιτύχουμε αυτό που ανέφερε ο ε, κύριος δηλαδή σύνολο 62 δισεκατομμυρίων ε, ε, δισεκατομμύρια επενδύσεις. Χρειαζόμαστε βεβαίως τις, προ... τις προσπάθειες και των κρατών μελών. Ε, λόγω των ε, προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε, ο στόχος αυτός δεν είναι εύκολο να επιτευχθεί. Γι' αυτό και θα ε, στη δομή του, μηχανισμού θα ε, ενταχθούν δύο δυνατότητες για τα κράτη-μέλη. Πρώτον, δεν ζητείται από τα κράτη-μέλη να χορηγούν επιδοτήσεις, απλώς εγγυήσεις από τον κρατικό τους προϋπολογισμό και αναλόγως της χώρας θα μιλούμε για ένα ποσοστό που θα ε, κατευθύνεται προς την εγγύηση και δεύτερον ότι η συμβολή ε, δεν θα ε, συνυπολογίζεται στον, στο έλλειμμα που προβλέπει το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Αυτό λοιπόν αποτελεί κίνητρο για τα κράτη-μέλη προκειμένου να συμβάλλουν. Και τέλος, κάτι που αφορά και τμήμα μιας ευρύτερης ε, προσπάθειας, στην οποία αναφέρθηκε και η κυρία Πρόεδρος, είναι το γεγονός ότι στην Επιτροπή Προϋπολογισμών αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις σχετικά με την παράταση της εντολής της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κάτι που θα έχει σημαντικότατες επιπτώσεις καθώς τμήμα του εξωτερικού επενδυτικού σχεδίου αφορά και την συνοχή μεταξύ της εξωτερικής εντολής της ΕΤΕΠ αλλά και της δικής μας πρωτοβουλίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Έχω δει ότι κάποιοι συνάδελφοι θέλουν ε, να, θέσουν κάποια ερωτήματα. Προσπαθώ να καταλάβω τι ακριβώς γίνεται και ίσως θα ήταν καλύτερα να κάνω εγώ κάποιε ερωτήσει πρώτα και μετά να δώσω το λόγο και στους ε, συναδέλφου. Μήπως έτσι καταλάβουμε καλύτερα τι ακριβώς είπατε. Αν κατάλαβα λοιπόν καλά, Από ό,τι κατάλαβα, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αϊφόρου Ανάπτυξης ε, έχει συμπεριλάβει δύο ε, ταμεία, την διευκόλυνση για την Αφρική και την επενδυτική διευκόλυνση για την ε, ευρωπαϊκή γειτονία πόσα από αυτά τα ποσά, τι από αυτά τα ποσά που αναφέρατε ήδη συμπεριλαμβάνονται στο, ε, στα ταμεία που υπάρχουν ε, και πόσο, ποιο είναι το συνολικό ποσό και για ποιο λόγο το κάνατε αυτό. Γιατί συγχωνεύσατε δύο μέσα σε ένα τώρα ξαφνικά. Ποια είναι η ιδέα πίσω από αυτό. Είναι ένα πρόβλημα ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η κατάσταση τώρα. Και ποιος είναι ο λόγος. Γιατί από ό,τι κατάλαβα δύο γενικές διευθύνσεις πρέπει να, να συνεργαστούν και αυτό είναι, ε, περιπλέκει κάπως τα πράγματα. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενθύσεων έτσι συμμετέχει καλύτερα. Δεν ξέρω ακριβώς για ποιο λόγο το κάνατε αυτό. Και είπατε ότι θα προκύψουν επίσης και κάποια χρήματα από χρηματοδότηση της Ένωσης. Εμείς αυτή τη στιγμή τι ε, προσφέρουμε. Και για να φτάσετε τα 3,35 δις που μας είπατε, τι χρειάζεστε ακόμα. Αυτά τα χρήματα, τα 3,35 δις προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή ε, αυτό είναι μόνο το 50% άρα υπολείπονται άλλα τόσα. Τώρα αν έχετε αυτή την ιδέα ότι είναι κάπως αυτό το εικονικό χρήμα το οποίο θα προέλθει από τα, ευρωπαϊκή, από τη, από τα ε, κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ως εγγύηση αλλά δεν είναι υπαρκτό χρήμα, δεν ξέρω αν είναι πάρα πολύ καλή ιδέα αυτό. Δεν κατάλαβα πάντως πολύ καλά για τι ποσά μας μιλήσατε, μήπως μπορείτε να μα τα αποσαφηνήσετε αυτά. Είπατε ότι θα γίνει και μια τεχνική συνεδρίαση την Παρασκευή, αλλά πρέπει και οι ευρωβουλευτές να μπορούν να το καταλάβουν. Μήπως ε, μπορείτε να μας πείτε λίγο περισσότερα πράγματα. Ίσως ε, να μας ε, ενημερώσετε σε σχέση με τα χρήματα που έχετε αυτή τη στιγμή, τι θα αλλάξει, για ποιο λόγο και ποια είναι η νέα πρόταση, γιατί μόνο το τεχνικό νομοθετικό κείμενο δεν μας αρκεί. Ίσως πρέπει να έχουμε και την τεχνική ενημέρωση με το ιστορικό που ε, δίνεται και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να καταλαβαίνουμε ακριβώς απολύτως ε, περί τίνος πρόκειται. Αν έχετε λοιπόν κάποιο έγγραφο επεξηγηματικό θα ήταν χρήσιμο. Είναι πιο πολιτικές ερωτήσεις που θα κάνω πιο μετά, αλλά για την ώρα είναι τεχνικές οι ερωτήσεις και θα αρκεστώ σε αυτές. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι εδώ μπαίνουμε σε μια συζήτηση πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Μόλις άκουσα τις δύο προσκεκλημένες ομιλήτριες και έχω πολλά σχόλια να κάνω. Πρώτον, η παρέμβαση στην Αφρική και στη γειτονία σκοπό έχει να δώσει προοπτικές ε, στον κόσμο επιτόπου για να τους αποτρέπει να φύγουν ε, και να ε, προσθεθούν στον ήδη μεγάλο αριθμό των μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το κατάλαβα. Δεύτερον, οι άνθρωποι που βρίσκονται εκεί όντως χρειάζονται προοπτική και θα ήθελα να συμφωνήσω με αυτό που είπε η Πρόεδρος, ε, τι στόχο προσπαθούμε να επιτύχουμε το Ταμείο για την Αηφόρο Ανάπτυξη θέλουμε να οδηγήσει σε αηφορία. Αν γίνει λοιπόν επένδυση πρέπει να γίνει κατά κύριο λόγο στο δημόσιο τομέα και στην επίσημη οικονομία. Όμως στην παραοικονομία, η παραοικονομία μήπως αυτομάτως θα επωφεληθεί και εκείνη κάποια ψυχουλάκια θα πάρει και η παραοικονομία τα ψυχουλάκια που θα πέσουν από την παρέμβαση στο δημόσιο τομέα. Το ερώτημα που θα ήθελα να θέσω όμως πιο συγκεκριμένα είναι το εξή. Μήπως είναι πιο πολύ περιοριστική αυτή η προσέγγιση, αν θέλουμε να υπάρξει αηφορία. Θα έπρεπε να προσανατολίζεται η αφορία αυτή στους στόχους της αηφόρου ανάπτυξης, ε, των ε, στόχων λοιπόν της χιλιετίας της Νέας Υόρκης. Δηλαδή στο τέλος θα πρέπει να υπάρχουν λιγότεροι φτωχοί γιατί έχω την εντύπωση ότι η παρέμβαση μπορεί να οδηγήσει σε περισσότερους πλούσιους και λιγότερους φτωχούς. Θα μπορούσαμε όμως ε, να έχουμε και λιγότερους πλούσιους και περισσότερους φτωχούς και θα μπορούσαμε να έχουμε και μια χαμένη προσπάθεια εντελώς. Εγώ λοιπόν αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι τι ακριβώς θα κάνουμε για να βγει ο κόσμος από την παραοικονομία Έχουμε στοχεύσει τα προγράμματα ε, προς αυτή την κατεύθυνση που είναι κατά τη γνώμη μου πάρα πολύ σημαντική, ειδικότερα στο πλαίσιο της ανάπτυξης. Ίσως είναι μια οδός που πρέπει επίσης να διερευνηθεί και θα ήθελα να συζητήσουμε και το θέμα κάπως ευρύτερα, όχι μόνο καθαρά, σε καθαρά οικομονικούς όρους. Ε, τουλάχιστον θα μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε και άλλα, άλλες διαστάσεις όταν θέτουμε το θέμα στις χώρες αυτές, για να μπορέσουμε να μειώσουμε τις ανισότητες ε, που βλέποντας μια σταθερότητα ε, η οικονομική τα αποτέλεσμα θα είναι και μεγαλύτερη παραγωγικότητα. Το να περάσουμε από την οικονομική ανάπτυξη πρέπει να οδηγεί πάντοτε σε μια ευρύτερη ανάπτυξη. Ε, αν θέλουμε λοιπόν με έξυπνες παρεμβάσεις στον κοινωνικό τομέα να προωθήσουμε την ε, οικονομική ανάπτυξη, νομίζω ότι θα προωθήσουμε έτσι έμεσα πολύ πιο αποτελεσματικά και την αηφόρο ανάπτυξη. Ε, επίσης, Μιλούμε εδώ για ένα νομοθετικό ε, κείμενο. Πρέπει να δώσουμε εμείς ε, τη συγκατάθεσή μας για να εκταμιευθούν κάποια ποσά και να, γίνουν κάποιες, να υπάρξουν κάποιες εγγυήσεις. Ο νομοθέτης ε, λοιπόν παρεμβαίνει μόνο στο περιθώριο. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι θα έχουμε διαφωτιστεί όσον αφορά την παρουσίαση των λογαριασμών. Μήπως μπορούμε να κάνουμε μία ενοποιημένη παρουσίαση όλων των παρεμβάσεων που στοχεύουν στην ανάπτυξη γιατί έχουμε τόσες πολλές παρεμβάσεις εκτός των ταμείων που καλύπτονται απευθείας από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε trust funds, Έχουμε συγχώνευση πολλών ταμείων, έχουμε τις ε, εγγυήσει και τις διευκολύνσεις. Νομίζω ότι είμαστε στη σωστή επιτροπή για να γνωρίσουμε λίγο περισσότερα πράγματα. Μήπως θα έπρεπε να υπάρξει μία δέσμευση στο πλαίσιο αυτής της νομοθετικής πρωτοβουλίας ε, για μία παρουσίαση ενοποιημένη των λογαριασμών για να υπάρχει μία παρακολούθηση ε, αρκετά πολιτική πέρα από την οικονομική. Εκτός από αυτά που μόλις είπα και τις ανησυχίες που εξέφρασα, συμφωνώ πάντως, είμαι μάλλον ε, σύμφωνος με όλα αυτά που ε, είπατε. Ε, έχω σκίσει κάποια κριτική, αλλά ελπίζω να είναι απλώς επικοδομητική. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συμφωνώ με τους προλαλήσαντες συναδέλφους, γιατί αυτά είναι σημαντικά ζητήματα. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε να αντιμετωπίσουμε την εξής κατάσταση. Βλέπουμε ότι η αιτιολόγηση για την δημιουργία νέων μέσων έχει να κάνει και πάλι με τη μετανάστευση και αυτό υπό το, την αποκαλούμενη ανάγκη να εξετάσουμε τα βασικά αίτια. Δεν είναι η πρώτη φορά, υπήρξαν ε, κι άλλα κι άλλα μέσα που τα αντιμετωπίσαμε κατά αυτόν τον τρόπο. Εμείς όμως είμαστε η μοναδική επιτροπή στην στο Ευρωπαϊκό ε, Κοινοβούλιο που πρέπει να εξασφαλίσει ότι ε, η αναπτυξιακή πολιτική όντως προωθεί την ανάπτυξη. Λιγότερη φτωχή θα πρέπει να υπάρχουν στην τελική ανάλυση, λιγότερη περιβαλλοντική καταστροφή πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχουν αυτοί οι μηχανισμοί που ε, ε, μετρούν, προσμετρούν τα αποτελέσματα σε σχέση με τους στόχους. Νομίζω ότι η ιδέα του κυρίου Γκέρενς είναι πάρα πολύ καλή. Ας τα συμπεριλάβουμε όλα αυτά ε, σε έναν κατάλογο ενοποιημένο για να δούμε ποιος είναι, ποιο είναι το αποτέλεσμα που μπορούμε να επιτύχουμε. Ε, ώστε να εξασφαλίσουμε το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα από αναπτυξιακής απόψεως. Πρέπει να καλέσουμε και τον ιδιωτικό τομέα. Πρέπει να παρέμβει σε μεγάλο βαθμό, δεν υπάρχει αμφιβολία. Αλλά έχουμε την καλύτερη εμπειρογνωμοσύνη για να κάνουμε κάτι τέτοιο. Ξέρουμε, είμαστε βέβαιοι ότι έχουμε ε, τους καλύτερους οργανισμούς ε, ως συμμετέχοντες. Εγώ δεν είμαι πεπισμένη για το ιστορικό της ΕΤΕΠ την προώθηση εξάλληψη τη της φτώχειας και άλλων αναπτύξεων στόχων. Παρακαλώ πείστε με λοιπόν, θέλω να πιστώ ότι υπάρχουν κοινωνικές δικλείδες ασφαλεία, ε, που λειτουργούν, που ε, ε, δουλεύουν πραγματικά και που θα μας βοηθήσουν να επιτύχουμε τους στόχους μας, όπως μόλις ακούσαμε. Επίσης θα ήθελα να πω ότι αυτή η ιδέα του Σάρλ Γκέρενς για την επένδυση στην κοινωνική προστασία, αν κατάλαβα καλά Σάρλ, είναι πραγματικά κάτι που θα πρέπει να σκεφτούμε. Δεν είμαι βέβαιη ότι η Παγκόσμια Τράπεζα έχει πολλή εμπειρογνωμοσύνη για το πώς τέτοιου είδους επένδυση κοινωνικής προστασίας για τους φτωχότερους σε αναπτυσσόμενες χώρες θα μπορούσε να οδηγήσει τον κόσμο ε, σε μια ε, πραγματική ε, ζωή που να έχει κάποια σημασία. Δεν ξέρω πώς αυτό είναι εφικτό στο πλαίσιο των υπαρχόντων μηχανισμών. Και τώρα, για το θέμα της παρακολούθησης, ακούσαμε, και αν κάνω λάθος ε, παρακαλώ Διορθώστε με αν δεν κατάλαβα καλά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα είναι στο Στρατηγικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου για την Αϊφόρο Ανάπτυξη, κατάλαβα καλά, τι είδου ε, αρμοδιότητες θα έχει αυτό το Στρατηγικό Συμβούλιο και ποιος ε, θα μπορεί να μοιράζεται αυτές τις πληροφορίες, ε, πόσο διαφανής είναι η επιλογή της στρατηγικής και, και οι στόχοι που τίθενται. Λοιπόν, πρώτα θα ακούσουμε τις απαντήσεις σε αυτές τις δύο ερωτήσεις, γιατί νομίζω ότι είναι καλύτερα έτσι από το να ακούμε όλες τις ερωτήσεις μαζί και μετά να χανόμαστε στην απάντηση. Λοιπόν, ακούσουμε πρώτα τις ε, ε, απαντήσεις σε αυτές τις δύο ερωτήσεις και μετά εσύ να κάνεις τις δυσκολότερε ερωτήσεις. Λοιπόν, να δώσω το λόγο τότε στις προσκεκλημένες μας απαντήσουν ε, στις ερωτήσεις που ετέθησαν από τους δύο συναδέλφους. Θα προσπαθήσω να εξηγήσω το πώς το βλέπω εγώ. Ποια είναι η επιπρόσθετη αξία αυτής ε, της πρωτοβουλίας. Είναι ότι για πρώτη φορά δημιουργούμε μία νέα εγγύηση, ένα νέο ταμείο εγγύησεων. Αυτό που προτείνουμε στον κανονισμό είναι να προσθεθεί το στοιχείο αυτό της ε, εκτάκτου ανάγκης ε, που δεν υπήρχε στο παρελθόν, γιατί μέχρι τώρα χρειαζόταν να ζητηθεί μια παρέκκληση από το ε, Ταμείο. Τώρα όμως τα χρήματα θα... Ε, κατευθύνονται καλύτερα γιατί θα υπάρχει ένα, μια βάση όπως ανέφερε η Καταρίνα. Θέλουμε λοιπόν να μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε ε, project σε τομείς υποδομής όπως υδατοδότηση, μεταφορές, ε, ε, υδροδότηση, μεταφορές κλπ με τρόπο που να ε, είναι επικερδής. Έτσι μπορούμε και στους φορολογούμενους να τα εξηγήσουμε καλύτερα. Προγράμματα τα οποία να μπορούν όντως να χρηματοδοτηθούν με κάποιο αποτέλεσμα. Θα τα βάλουμε τότε σε μία πύλη, θα σας τα εξηγήσουμε, θα υπάρξει ένα στρατηγικό συμβούλιο, ένα επιχειρησιακό συμβούλιο ε, ε, όλα αυτά θα είναι πολύ σαφώς καθορισμένα και θα μπορούμε να ξέρουμε τι ακριβώς είναι δυνατό να χρηματοδοτηθεί. Θα υπάρχει διαφάνεια, θα υπάρχει λογοδοσία και είναι κάτι το οποίο θα λειτουργήσει. Να χρησιμοποιούνται οι επιδοτήσεις για αυτά τα προγράμματα για την υγεία, την εκπαίδευση, την κοινωνική προστασία που αναφέρατε κι εσείς τα οποία θα τα χρηματοδοτήσουμε όντως με επιδοτήσεις, με το κοινωνικό κομμάτι της ανάπτυξης που αναφέρατε, δηλαδή την αντιμετώπιση της φτώχειας, των ανισοτήτων κλπ. Αυτά εν η μακροπρόθεσμη αηφορία, η μακροπρόθεσμη απασχόληση ε, θέσεις εργασίας ε, και αντιμετώπιση των βασικών αιτιών ε, της φτώχειας και της ε, μετατόπισης των ε, πληθυσμών, της μετανάστευσης. Αυτή είναι η ομορφιά του σχεδίου μας. Τώρα, όσον αφορά τη χρηματοδότηση, θα σας δώσουμε βεβαίως την τεχνική ενημέρωση και όλες τις πληροφορίες. Όπως είπα, θα προέλθει από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης και όχι από τον προϋπολογισμό 3,2 συνολικά και από τον ενωσιακό προϋπολογισμό ε, θα υπάρξουν κάποια στοιχεία από το αποθεματικό και θα σας δώσουμε και έναν κατάλογο ε, και τον προγραμματισμό για να δείτε από ποια γραμμή του προϋπολογισμού θα βγει το κάθε ποσό. Αυτά λοιπόν για τον αναπτυξιακό αντίκτυπο, για το ρόλο τώρα της ΕΤΕΠ. Βεβαίως ε, και θα υπάρξει ρόλος για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, στρατηγικός ρόλος. Εμείς θέλουμε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να είναι εκεί ως παρατηρητής και θα ήθελα να σας πω ε, βεβαίως ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα είναι ένα από τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα που θα εφαρμόσουν το ε, σχέδιο αυτό, όπως είπε και η Καταρίνα. Ευχαριστώ. Um, thank you. Um, just to uh, compliment uh, για να συμπληρώσω ορισμένα σημεία, όπως είπε και η Μαριέτα, υπάρχει αυτό το νέο χρήμα που προαναφέρουμε, που προέρχεται από το προϋπολογισμό του της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή 750 εκατομμύρια συν 750 και μαζί με τα 3,5. Μας ρωτήσετε όμως γιατί γίνεται αυτό. Και η Μαριέτα είπε ότι ο συνολικός στόχος είναι αυτός που γνωρίζετε. Ένας από τους λόγους, είπε, όπως είπε και ο κύριος Γκέρενς, είναι ότι θα πρέπει να έχουμε ένα συνδυασμό των μέτρων για την αναπτυξιακή βοήθεια. Ίσως δεν είναι ένας εύσχημος τρόπος γιατί τα πράγματα ε, εξελίσσονται στην Ευρώπη κατά κατακαιρματισμένο τρόπο πολλές φορές. Εμείς θέλουμε να υπάρχει μία συνεκτική ομπρέλα, στο το πω έτσι. Και αυτό μέσα στα πλαίσια και των εγγυήσεων, επί των οποίων θα νομοθετήσετε, σε σχέση με ένα δηλαδή μόρφωμα. Υπάρχουν δύο μέσα αλλά χρησιμοποιούμε ένα ενιαίο μέσο για να τα εντάξουμε όλα. Δεν είναι ιδεατός αυτός ο τρόπος, αλλά βραχυχρόνια αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να υπάρξει συνοχή στις αναπτυξιακές μας προσπάθειες για να αντιμετωπίσουμε δραστικά το θέμα της μετανάστευσης. Δεν το κάνουμε ε, ολιστικά, προσπαθούμε να το κάνουμε κατά βήμα για να υπάρχει κάποια συνοχή, γιατί ε, αισθανόμαστε ακριβώς το ίδιο όπως και εσείς, γιατί έχουμε τα διάφορα τα καταπιστεύματα, τα διάφορα μέσα, εργαλειοθήκες και ούτω καθεξής. Γι' αυτό θέλουμε να υπάρχει αυτή η τακτική της συμπερίληψης, ε, δηλαδή με τις δικές μας επιδοτήσεις να αντιμετωπιστούν και οι δανειοδοτήσεις, έτσι ώστε να υπάρξει συνολικά και ένα ταμείο εγγύησαν έτσι ώστε να συμπεριληφθεί και ο ιδιωτικός τομέας. Όπως είπε και η κυρία Χαουτάλα, θέλουμε ο ιδιωτικός τομέας να μπορέσει να συνεισφέρει στους αναπτυξιακούς στόχους, κάτι το οποίο δεν έχει γίνει ακόμα, διότι είναι δύσκολο και την Παρασκευή όταν γίνουν οι συζητήσεις τεχνικής υφής θα καταλάβετε πόσο δύσκολο είναι έμπρακτα. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να ε, βάλουμε και τα νέα στοιχεία, δηλαδή τον ε, ιδιωτικό τομέα και την συνοχή ως προς τα μέσα. Για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε σωστά με τους εταίρους σε σχέση με την ε, υπόγεια οικονομία και την ε, κοινωνική πτυχή. Αυτές είναι οι μεταρρυθμίσεις που αφορούν τον πυλώνα υπαριθμών 3 και υπάρχει και ο δεύτερος πυλώνας για την τεχνική βοήθεια. γιατί η υπόγεια οικονομία δεν μπορεί να βγει στην επιφάνεια τόσο εύκολα. Είτε πρόκειται για, το, για μια τράπεζα του Περού, είτε για άλλα μέσα έτσι ώστε να έχουμε την ένταξη της υπόγειας οικονομίας στην επίσημη. Ε, Ελπίζουμε λοιπόν να συνδυάσουμε και τα δύο. Ε, δύο ερωτήσεις, ε, Πατρίσια Τόια και Νόρπερτ Νόιζερ. Μετά θα περάσουμε στους δύο επόμενους ομιλητές. Εκτιμώ τις προσπάθειές σας και όλα τα συστατικά μου φαίνονται σωστά για την ε, υπόγεια οικονομία. Όμως, παρά τα συστατικά, θεωρώ ότι η συνταγή δεν είναι καλή. Θα ήθελα να κάνω ορισμένες παρατηρήσεις επικοδομητικά. Είτε θα κάνουμε όμως ένα ποιοτικό άλμα για την ανάπτυξη της Αφρικής, Διαφορετικά βελτιώνουμε κάπως τις πολιτικές, τις μέχρι τώρα πολιτικές, χωρίς να ξέρουμε τι συμβαίνει πραγματικά. Οι αναπτυξιακές μας πολιτικές ήταν στοχοθετημένες. Σήμερα όμως θα πρέπει να δώσουμε μία τελική μορφή σε αυτές τις πολιτικές, γιατί έχει εξελιχθεί η κατάσταση. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και το μεταναστευτικό, το οποίο όλο ένα και διονγκώνεται. Γιατί υπάρχουν και ολέθριες συνέπειες κοινωνικής υφής. Άρα είτε θα κάνουμε κάτι το καινοτόμο ή δεν ξέρω πώς θα αντιμετωπίσουμε τη μετανάστευση. Εάν ε, δεν θεωρήσουμε ότι αυτό είναι προτεραιότητα, τότε είμαστε εκτός ε, ιστορικού πλαισίου. Στη χώρα μου φτάνουν σε δύο μέρες το Σαββατοκυριακό. Το, ο αντίστοιχος φτάνει ο αντίστοιχος αριθμός ε, των παρεπιδημούντων στο καλέ. Αν ο καιρός είναι καλός τα Σαββατοκύριακα. Άρα είτε θα δοθεί μία απάντηση υποδοχής, αλλά εάν δεν ξέρουμε τι συμβαίνει στην άλλη πλευρά της Μεσογείου, τότε δεν αντιμετωπίζουμε τίποτα. Δεν χρειάζεται να προσθέσουμε την εγγύηση. Είτε λοιπόν θα δώσουμε μία νέα διάσταση στο ζήτημα, γιατί είναι ένα από τα λίγα χαρτιά που έχουμε στο χέρι μας ή δεν, ε, μπορούμε να καταφέρουμε τίποτα. Καταλαβαίνω το θέμα της συνοχής. Αν έχουμε όμως το, το Ταμείο γειτονία και το Ταμείο Αγγίσεων, πώς θα μπορέσουμε να τα βάλουμε μαζί όλα αυτά, να τα εντάξουμε το ένα μέσα στο άλλο. Υπάρχει και το κοινωνικό και η υπόγεια οικονομία και δυστυχώς όλα αυτά θα αποδομηθούν. Γι' αυτό δεν πρέπει να καταστρέψουμε αυτό το πλαίσιο πριν δημιουργηθεί. Γιατί θέλουμε να συμμετάσχει και η κοινωνία των πολιτών. Δεν πρέπει όμως να κατακαιρματίσουμε αυτή την προσπάθεια. Καταλαβαίνετε ότι η Ιταλία είμαστε, είναι η εμπροστοφυλακή. Μπορεί να είναι και η Ελλάδα, οι βαλκανικές ε, χώρες και ούτω καθεξής. Αλλά εγώ μιλάω για την Ευρώπη. Μας ενδιαφέρουν τα σχέδια, αλλά όχι μεμονωμένα. Μιλάμε για στρατηγική επιτροπή, ε, υποεπιτροπές, ε, υποδιαρθρώσεις. Αυτό που έχει σημασία είναι η Επιτροπή να αναλάβει τις ευθύνες ε, της. Μην κάνετε εξωτερικές αναθέσεις για όλα. Και σας το λέω με κάθε ειλικρίνεια. Εσείς πρέπει να προβάλλετε σχέδια και προγράμματα με τις ενδιαφερόμενες χώρες. Μην κάνετε εξωτερικές αναθέσεις. Είναι πολύ εύκολο κάτι τέτοιο. Θα πρέπει να υπάρχει μία πολιτική πλαισίωση. Δεν μπορείτε να μιλάτε για ομπρέλες, για πλαισιώσεις. Θα πρέπει να μας πείτε τι μπορεί να γίνει μεταξύ Ευρώπης και της χώρας Χ. ποιο πρόγραμμα θα προβάλλεται για συγκεκριμένες χώρες, ε, τι θα γίνει στον τομέα των υδάτων, της ενέργειας, της αγροτικής οικονομίας. Δηλαδή, ας ε, φτάσουμε σε απτά προγράμματα. Καταλαβαίνω τις δυσκολίες, αλλά ας υπάρχουν ορισμένες εγγυήσεις, μίνιμουμ εγγυήσεις. Δηλαδή, ποιο είναι το απτό πρόγραμμα που έχετε κατά νου και ποιες είναι οι δεσμεύσει σας και επιτοπίως. Γιατί φυσικά υποδεχόμαστε τους πρόσφυγες, αλλά ποιες είναι οι υποδομές για να εντάξουμε ας πούμε τα ορφανά παιδιά που έχουν διασχίσει τη Μεσόγειο πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχει μία ε, απλή στοχοθέτηση. Νόρμπερτ Νόιζερ. Λυπάμαι. Ο Τσάρλς Κιόρεν μόλις μίλησε για τους κοινού θνητούς. Και είμαι κι εγώ ένας από αυτούς τους ε, κοινού και δυστυχώς δεν κατάλαβα την προσέγγιση της Κομισιόν. Αν πάρουμε το 1,5 δις για περαιτέρω μέτρα, ιδίως για τους πρόσφυγες. Αυτό σημαίνει, ή τουλάχιστον εγώ έτσι το εκλαμβάνω, ότι πρόκειται για ένα θετικό μέτρο. Αν όμω ταυτόχρονα χρειαζόμαστε νέα εργαλεία και νέα μέσα, σημαίνει ότι είναι και μια παραδοχή ότι τα παλιά μας εργαλεία δεν έφεραν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Άρα γιατί χρειαζόμαστε τώρα αυτό το νέο μέσο. Επίση, γιατί χρειαζόμαστε τώρα εγγύησει. Παλιότερα δηλαδή δεν υπήρχαν εγγύησει όσον αφορά την αναπτυξιακή ε, βοήθεια. Τέλο, μα υπόθηκε ότι ε, ο, το κοινοβούλιο θα έχει ένα ρόλο παρατηρητή. Με συγχωρείτε πολύ, αλλά αν ο ρόλος που μα επιφυλάσσεται είναι εκείνο του παρατηρητή, τότε μπορούμε να το εγκαταλείψουμε από τώρα το θέμα. Θα προσπαθήσω να απαντήσω εντάχει αυτό που θέλει η Επιτροπή είναι να πλαισιώσει και να εντάξει όλες τις πρωτοβουλίες υπό μία σκέπη. Γι' αυτό θέλουμε να υπάρχει συνοχή και συνέπεια στις πολιτικές μας. Εμείς δεν υπε... υπεκφεύγουμε των ευθυνών μας. Η Επιτροπή φέρει την ευθύνη. Εμείς θα αναλάβουμε τη γραμματιακή υποστήριξη, το One Stop Shop και εμείς θα είμαστε υπεύθυνοι ως Κομισιόν. Θα προσπαθήσουμε επίσης να εντάξουμε τα προγράμματα ανάλογα με τις θεματικές ανάγκες, τις γεωγραφικές ανάγκες, περιφερειακές, τομεακές και ούτω καθεξής. Δηλαδή θα λάβουμε υπόψη το στρατηγικό ρόλο αυτού του στρατηγικού συμβουλίου που θα ασχοληθεί με τις προτεραιότητες. Γι' αυτό είναι και πάρα πολύ σημαντική η συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρατηγικό Συμβούλιο. Εσείς είσαστε ο κοινός νομοθέτης, ο συνομοθέτης, δεν θα σας πω τι να κάνετε, αλλά θα θέλαμε να συμμετάσχετε ενεργά. Ε, δεν μπορεί να γίνει τίποτα χωρίς τη συμμετοχή σας. Και αυτό προσπαθώ να σας πω για την άμεση συμμετοχή σας και στο Στρατηγικό Συμβούλιο. όλα αυτά μέσα στα πλαίσια της συνεκτικής ε, πολιτικής. Εντάχει, θα ήθελα να πω στην ε, Ιταλίδα Ευρωβουλευτή, ε, μας ε, μιλήσατε για τα επιμέρους ε, θέματα σε σχέση με την εγγύηση και την πολιτική ανάμιξης και ένταξης. Υπάρχουν όμως και διμερεί προγράμματα με τις χώρες αυτές όπου υπάρχει μια πολιτική διαλόγου. Θέλουμε λοιπόν να δημιουργήσουμε ένα μηχανισμό ο οποίος να συμβαδίζει με την διμερεί βοήθεια Δηλαδή αυτό είναι ένας υποτομέας. Νομίζω ότι στις περιφέρειες είναι απόλυτα σαφές ποια κονδύλια πάνε πού ή ποια ταμεία απευθύνονται σε ποιον και πού μπορεί να υποβάλει αίτηση κανείς, γιατί κάθε φορά που το συζητάμε Μιλάμε για τις γυναίκες, για τη φτώχεια, αλλά θα θέλαμε να ξέρουμε ποια είναι αυτά τα χρηματοδοτικά μέσα. Ας ε, μην ε, ε, λέμε ότι είναι κάτι που δεν είναι η χάιντι. Ναι, μιλάμε για συνοχή και για τη νέα πλαισίωση. Νομίζω ότι θα πρέπει να σταματήσουμε ίσως, να βοηθήσουμε να σταματήσει η μετανάστευση. Δηλαδή, ας ασχοληθούμε με τη φτώχεια και τις ανισότητες και όχι τόσο με τη μετανάστευση καθεαυτή. Γιατί φτάνουμε σε εσφαλμένα συμπεράσματα. Δηλαδή η ανάπτυξη δεν θα σταματήσει τη μετανάστευση. Ε, είναι βεβαιασμένα τα πράγματα έτσι όπως τα θέτεται. να πω ότι αυτό που θέλουμε είναι ως γενικές διευθύνσεις να αξιοποιήσουμε όλες τις δυνατότητές μας, να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια προκειμένου να ενισχύσουμε την μακροπρόθεσμη και βιώσιμη ανάπτυξη στις χώρες εταίρους. Αυτό είναι ο κύριος στόχος και από εκεί και πέρα βεβαίως δεν χάνουμε από τον προσανατολισμό μας και τα υπόλοιπα που αναφέρατε. Πρόεδρος, να, πάρουμε τώρα, να πάμε τώρα στους άλλους ομιλητές. Το Συμβούλιο ε, που έχει συζητήσει σε ε, πολύ μεγάλο βαθμό και σε πολύ μεγάλη έκταξη το ζήτημα της μετανάστασης. Περνάμε τώρα στο δεύτερο τμήμα. Ο κύριος Νταυγκίλοβιτς από την ΕΤΕΠ πρώτα, στη συνέχεια Νατάλια Αλόνσο από την Oxfam. Κύριε Νταγκυλόβιτ, έχετε τον λόγο. Νικολάη, αν μου επιτρέπετε. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ που προσπαθήσατε να προφέρετε σωστά το όνομά μου. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκλησή σας να παραστώ εδώ στην Επιτροπή σας. Είναι η πρώτη μου φορά που βρίσκομαι στην Επιτροπή Ανάπτυξης. Εμάς μας ενδιαφέρει να υπάρχει ένας καλός διάλογος μαζί σας. Ε, είναι ήδη πέντε το απόγευμα, αλλά θέλω να σας υπενθυμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αποτελεί σημαντικό παράγοντα της ε, ε, Ευρωπαϊκής Αναπτυξιακής Βοήθειας και ο ρόλος μας διευρύνεται χρόνο με το χρόνο. Κάτι που αποδεικνύει και το γεγονός ότι ο ρόλος που έχει ανατεθεί στην ΕΤΕΠ δεν είναι απλά και μόνο να κάνει αναπτυξιακή βοήθεια γιατί θεωρούμε ότι είναι ενδιαφέρουσα, αλλά επειδή κάτι τέτοιο πηγάζει από τις ευρωπαϊκές συνθήκες. Μπορούμε, μπορώ να σας πω ε, τι κάνουμε στην Ανατολική Αφρική για τις συνθήκες υγιεινής ή για την γυναικεία επιχειρηματικότητα δεν θα το κάνω γιατί είναι ήδη αργά, αλλά θα μπορούσαμε να, διοργανώσουμε ένα σεμινάριο για τους υπαλλήλου αλλά και τους ευρωβουλευτές του Κοινοβουλίου προκειμένου να σας δείξουμε τι κάνουμε και πόσες προσπάθειες καταβάλουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Επίσης, πρέπει να σας πω ότι είμαστε, η Κομισιόν είναι πολύ περήφανη για την ε, πρότασή της αυτή, η οποία κατέστη δυνατή να καταρτιστεί ε, υπό πολύ ψηλή ε, πίεση γιατί κάθε μέρα βλέπουμε στις ειδήσει τι συμβαίνει στις ακτές της Μεσογείου και εγώ συμφωνώ πολύ ε, με αυτό που είπε η κυρία Τιστόγια όσον αφορά τη μετανάστευση. Δεν θα πρέπει να κάνουμε λοιπόν αυτήν την τεχνητή συζήτηση για διάφορες έννοιες. Αντιθέτως, νομίζω ότι η Κομισιόν έχει καταβάλει πολύ μεγάλες προσπάθειες προκειμένου να αναπτυχθούν σύγχρονα μέσα που δίνουν τη δυνατότητα κινητοποίησης και αξιοποίησης ε, οικονομικών πόρων που βρίσκονται σε έλλειψη βεβαίω, δεν χρειάζεται να σα το υπενθυμίσω αυτό. Και εμεί ω ΕΤΕΠ συνεργαζόμαστε και με την Κομισιόν αλλά και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να, καταφέρουμε να επιτύχουμε ακριβώ αυτόν τον στόχο. Εμεί ε, έχουμε ε... μηχανισμού του οποίου έχουμε αξιοποιήσει και που είναι βεβαίως διαφορετικοί, αλλά έχουν το ίδιο κοινό στοιχείο. Τους τρεις πυλώνες και την αιρεσιμότητα. Είναι σημαντικό να εξετάσει κανείς αυτόν τον πρώτο και τον τρίτο ιδίω πυλώνα. Επίσης, αυτό που μας ενδιαφέρει πολύ είναι όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να μπορούν να αξιοποιήσουν στο έπακρον τις δυνατότητές τους προκειμένου να συμβάλλουν ε, στην επιτυχία του σχεδίου αυτού. Και νομίζω ότι μέσω των εργασιών στο Συμβούλιο καταφέραμε κατά κάποιον τρόπο να αποκτήσουμε και μια σαφέστερη εικόνα για το πώς θα μπορούσε να τεθεί στην πράξη, να υλοποιηθεί στην πράξη αυτό το σχέδιο. Και εμείς από την πλευρά μας συμβάλλουμε ε, όσον αφορά την, τη διάσταση της χρηματοδότησης και της πίστης ε, προκειμένου το σχέδιο να καταστεί λειτουργικό το συντομότερο δυνατό. Επίσης, θέλω να πω ότι φυσικά θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι και τα άλλα μέσα και εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας, και εδώ η ΕΤΕΠ, όπως ίσως έχετε ακούσει, η ΕΤΕΠ λοιπόν έχει προτείνει και έχει λάβει την έγκριση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Ιούνιο μια πρωτοβουλία που ε, λέγεται ε, «Πρωτοβουλία για την ανθεκτικότητα των, ε, της ε, Ανατολικής Γειτονίας και των Νοτίων Βαλκανίων προκειμένου να ενισχυθούν οι προσπάθειές μας και οι ενέργειές μας στις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο από τη μετανάστευση. Και χωρί να μπω σε πολλέ λεπτομέρειε σχετικά με αυτή την πρωτοβουλία, θα ήθελα κάποια στιγμή να έχουμε την ε, δυνατότητα να σα την παρουσιάσουμε, γιατί νομίζουμε ότι είναι πολύ ε, ενδιαφέρουσα και αυτή. Για μα λοιπόν αυτό που ήταν σημαντικό ήταν να εξασφαλίσουμε ότι όλα τα εργαλεία θα μπορούν να ε, τίθενται σε λειτουργία και να αξιοποιούνται ταυτόχρονα και από κοινού, χωρί να υπάρχουν διάφορα στρώματα γραφειοκρατία που θα δυσκολεύουν το έργο μας. Και νομίζω ότι η Κομισιόν έχει καταφέρει ε, να κινηθεί ακριβώς σε αυτή την κατεύθυνση. Συμπερασματικά λοιπόν, νομίζω ότι η πρόταση που θα λάβετε από το Συμβούλιο θα είναι πολύ καλή. Δεν μπορώ βεβαίω εγώ να σα το υποσχεθώ αυτό, γιατί δεν είμαστε εμεί ο νομοθέτη. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω ότι πρόκειται για μία δέσμη μέτρων η οποία κινείται στη σωστή κατεύθυνση και που νομίζω ότι ε, ε, είναι ένα νομοθέτημα, μια δέσμη μέτρων που θα προταθεί και όπου εμεί θα έχουμε ε, πολύ, μεγάλη, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πολύ μεγάλη χαρά να συμμετάσχουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, λέει πρόεδρος. Η Νατάλια Αλόνσο από την Oxfam έχει τον λόγο και μπορούμε να ακούσουμε στη συνέχεια και τη γνώμη της Plan International. Ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να μοιραστούμε μαζί σας τις ανησυχίες της κοινωνίας των πολιτών. Εμείς χαιρετίζουμε το ενδιαφέρον της Κομισιόν να ε, αναπτύξει αυτήν την επενδυτική πρωτοβουλία, ωστόσο θα θέλαμε να διδαχθούμε και από τα, τις εμπειρίες, τις θετικές και αρνητικές εμπειρίες που έχουμε συλλέξει στο παρελθόν. Θα ήθελα λοιπόν να επικεντρωθώ σε κάποια βασικά ζητήματα και ενδεχομένως να σας υποβάλω και κάποιες συστάσεις στο τέλος. Ο στόχος λοιπόν μιας τέτοιας πρωτοβουλίας όπως, αυτό το, όπως είναι αυτό το εξωτερικό επενδυτικό σχέδιο θα ήθελα να μιλήσω για το πρόβλημα, το κυρίως πρόβλημα και στη συνέχεια να σας δώσω ε, πώς, ε, κάποιες συστάσεις για το πώς μπορούν οι επενδύσεις να αξιοποιηθούν για την εγκαταπολέμηση της φτώχειας και των ανισοτήτων. Πρώτον, ποιο είναι το πρόβλημα και ποια είναι η λύση. Να ε, επανέλθουμε λιγάκι στην βασική έννοια. Η μετανάστευση είναι πρόβλημα. Εμείς δεν πιστεύουμε ότι η μετανάστευση είναι πρόβλημα. Εδώ και χιλιετίες οι άνθρωποι μετακινούνται και μεταναστεύουν για διάφορους λόγους. Είναι σύνθετο το, το φαινόμενο, αλλά χρειάζεται διαχείριση. Η καλή του διαχείριση δε μπορεί να αποβεί αμοιβαία αποφελής για όλες τις πλευρές. Μάλιστα η μετανάστευση μπορεί να συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη, ιδίως όταν συνοδεύεται από κατάλληλες λύσεις. Το ερώτημα λοιπόν ε, για μας, η απάντηση μάλλον είναι ότι ε, η μετανάστευση δεν είναι πρόβλημα. Μα αν η μετανάστευση ή δεν είναι πρόβλημα, τότε γιατί το εξωτερικό επενδυτικό σχέδιο προσπαθεί να αντιμετωπίσει τα ε, γενεσιουργά αίτια της μετανάστευσης. Εμείς λοιπόν αναγνωρίζουμε αυτόν τον θετικό συσχετισμό ανάμεσα στη μετανάστευση και την ανάπτυξη και νομίζουμε ότι αυτή η πρωτοβουλία θα έπρεπε να επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση του εκτοπισμού γιατί λοιπόν οι άνθρωποι εγκαταλείπουν τις αιστείες τους. Θα έπρεπε Γι' αυτό το λόγο να επικεντρωθούμε στην ε, βελτίωση της διακυβέρνησης και στην καταπολέμηση των ανισοτήτων και να δοθεί η δυνατότητα στους πολίτες να ζητούν οι κυβερνήσεις τους να λογοδοτούν. Γι' αυτό και θεωρούμε ότι το εξωτερικό επενδυτικό σχέδιο θα έπρεπε να ε, συνδέει την διαχείριση της μετανάστευσης με την επίτευξη των στόχων για την οικονομική ανάπτυξη και να εξασφαλίζει τα δικαιώματα των δικαιούχων και όχι να αποτελεί έναν μοχλό άσκησης εξωτερικής πολιτικής. Αυτό ως προς το πρώτο ερώτημα. Ως προς το δεύτερο ερώτημα. Ναι, πράγματι, χρειάζεται να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Αλλά η ανάπτυξη δημιουργεί αυτόματα νέες θέσεις εργασίας. Γνωρίζουμε ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Το έχουμε δει στην Ευρώπη και σε αναπτυσσόμενες χώρες. Η Νιγηρία, για παράδειγμα, έχει ρυθμούς ανάπτυξης 5% τα τελευταία χρόνια. Ξέρετε όμως κάτι. Η φτώχεια έχει αυξηθεί από το 54% στο 70%. Άρα η οικονομική ανάπτυξη δεν αποτελεί έναν μοχλό που αυτόματα οδηγεί στη μείωση της φτώχειας ή στην αύξηση των θέσεων εργασίας. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια διαφορετική προσέγγιση για να αντιμετωπιστεί η φτώχεια και οι ανισότητε. Γι' αυτό και θεωρούμε ότι χρειάζεται μια εντελώ διαφορετική λογική όσον αφορά τι επενδύσει. Πώ μπορούμε λοιπόν να καταστήσουμε αυτή την πρόταση για τι επενδύσει ώστε αυτή να αντιμετωπίζει πραγματικά τι ανισότητε και τη φτώχεια. Πρώτον, το ζήτημα του blending, τη συγχώνευση. Κάθε ευρώ που κατευθύνεται στην συγχώνευση με την, ε, με την ε, δημόσια εκπαίδευση είναι ευρώ που χάνεται από τις άμεσες επενδύσεις. Γι' αυτό και χρειάζεται να ε, αποδεικνύεται κάθε φορά η συμπληρωματικότητα. Άρα, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι κάθε ευρώ που θα κατευθύνεται θα βρίσκει τον στόχο για τον οποίο έχει διατεθεί. Δεύτερον, οι προσπάθειες της ΕΤΕΠ στο πλαίσιο του blending, της συγχώνευσης, γίνεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ποια είναι λοιπόν τα διδάγματα που έχουν αντληθεί από τα ε, συστήματα και τους μηχανισμούς του, του Έχουμε διδαχθεί, έχουμε αντλήσει διδάγματα και πώς αυτή η συμπληρωματικότητα μπορεί να αποδειχθεί σε κάθε ξεχωριστή περίπτωση. Η σύσταση η δική μας λοιπόν είναι πώς μπορούν τα διδάγματα να ενσωματωθούν στο επενδυτικό σχέδιο. Το τρίτο στοιχείο και χαίρομαι πολύ για τις ε, εγγυήσεις και τις ασφαλιστικές δικλίδες που μας ανέφεραν όσον αφορά τα, τα κοινωνικά ζητήματα ή το περιβάλλον ή κομισιόν. Υπάρχουν λοιπόν ε, κίνδυνοι που, που ενέχονται όταν κανείς ε, αναμειγνύει δημόσιους και ιδιωτικούς οικονομικούς πόρους. Ε, σε διάφορους δείκτες, διάφοροι δείκτες που ε, φαίνονται να ευημερούν, να το πω έτσι, συνδέονται με την καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και αυτό αφορά κυρίως τις πολυεθνικές αλλά και τη δραστηριότητα εταιριών σε αναπτυσσόμενες χώρες όπου δεν υπάρχει συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο που να διέπει τη λειτουργία τους. Άρα, το ερώτημα που μας απασχολεί εμάς είναι πώς θα μπορούσε να ενισχυθεί η λογοδοσία του σχεδίου αυτού, πώς μπορούν να αυστηροποιηθούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και πώς μπορεί ε, να εξασφαλιστεί η ανάληψη ευθύνης από τις ίδιες τις τράπεζες. Να υπάρχει δηλαδή, για παράδειγμα, μια πρόβλεψη οι εταιρείε που θα είναι επιλέξιμες να μην φοροαποφεύγουν και να ανταποκρίνονται στις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Επίσης, πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι η χρηματοδότηση θα είναι διαφανής. Έχουμε συζητήσει για το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ε, το οποίο πρέπει και μπορεί να συμβάλλει στη διαφάνεια αυτού του νέου εργαλείου. Θέλουμε να ενισχυθεί η αξιολόγηση και η παρακολούθηση προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι το εργαλείο αυτό, το σχέδιο αυτό θα αποφέρει τα μέγιστα δυνατά ωφέλη. Όσον αφορά την υποβολή εκθέσεων, υπάρχει και ένα ζήτημα διαθεσιμότητας και διαφάνειας των δεδομένων και πώς αυτά επηρεάζουν τη ζωή των ανθρώπων και την εξάλληψη της φτώχειας. Έχουμε και εδώ λοιπόν κάποιες συστάσεις. Να... Θα ήθελα να μοιραστώ το χρόνο μου με τον Αλεξάνδρ Μακρόφ προκειμένου να σας μιλήσει ε, για αυτό το θέμα. Ε, η πρόεδρος λέει, μπορείτε να πείτε δύο λόγια αλλά να ξέρετε ότι έχετε ήδη ε, ε, ε πάρει όλο το χρόνο σας. Έχουμε ακούσει πολλά για το ρόλο σας ε, στην ε, εφαρμογή ε, του σχεδίου και είναι γεγονός ότι οι γενικές γραμμές ε, συχνά ε, μειώνεται ο χώρος ε, για τους πολίτες της αναπτυσσόμενες χώρες, είναι μειωμένος μάλλον αυτός ο χώρος. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι πρέπει να ενδυναμώσουμε τους πολίτες, να συνεργαστούν με τις κυβερνήσεις, να έχουν κοινέ προτεραιότητες για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων και της φτώχειας, να εξασφαλίσουμε λοιπόν ότι ο κανόνας της κοινωνίας των πολιτών και του χώρου για τους πολίτες ε, είναι όντως, ε, έχει όντως ληφθεί υπόψη σε ε, ό,τι κάνουμε. Πρέπει να εξασφαλίσουμε επιτόπου ότι η κοινωνία των πολιτών συμμετέχει στις συζητήσεις και αυτό είναι κάτι το οποίο μας απασχολούσε πάρα πολύ όταν μας παρουσιάστηκε το σχέδιο στα τέλη Αυγούστου γιατί ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών δεν ήταν αρκετά σημαντικός και ίσως ε, να είναι και ο λόγος που υπάρχει ένας τέτοιου είδος κανόνας, ε, γιατί σας αναφερθήκατε για το ρόλο του, στον ρόλο του Ευρωπαϊκού ε, Κοινοβουλίου, αλλά θα είναι σημαντικό να αναφέρονται και η, και η κοινωνία των πολιτών και οι πολίτες των χωρών εταίρων να συμμετέχουν σε εξίσου σημαντικό βαθμό. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Χάουτελα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, απλώς ε, για να σας πω, είναι πάρα πολύ καλό το ότι κάνουμε αυτή την τόσο σημαντική συζήτηση αυτή τη στιγμή, γιατί ακόμα τα πάντα είναι δυνατά. Μπορούμε τα πάντα να τα βελτιώσουμε ακόμη. Ακούσαμε τώρα από την Oxfam ότι το πρόβλημα δεν είναι ήδη, δεν είναι ουσιαστικά πρόβλημα, ε, και ότι η λύση δεν αποτελεί ουσιαστικά λύση στο πρόβλημα αυτό που δεν είναι πρόβλημα. Οπότε μπορούμε να αρχίσουμε να συζητούμε πώς θα ε, μετατρέψουμε όλη αυτή την κατάσταση σε ένα πραγματικό μέσο για την αντιμετώπιση της φτώχειας και των ανισοτήτων για να μπορέσει ο κόσμος ε, να ζει μια αξιοπρεπή ζωή σεβόμενος στο περιβάλλον. Θα ήθελα απλώς να σας πω ότι αν η κλιματική αλλαγή ε, συνεχιστεί όπως εξελίσσεται ως τώρα, έχουμε δει μόνο 1% του αριθμού των ε, προσφύγων που ε, θα δούμε αν ε, εξελιχθεί πολύ άσχημα η περιβαλλοντική καταστροφή. Πρέπει λοιπόν να σταματήσουμε να μιλούμε απλώς για μετανάστευση, αλλά να αντιμετωπίσουμε και την ενδεχόμενη κλιματική, την κλιματική αλλαγή και την ενδεχόμενη περιβαλλοντική καταστροφή που αυτή θα σημαίνει, γιατί όταν θα φτάσει γιατί έχει φτάσει η στιγμή να συζητήσουμε ε, το πραγματικό νόημα όλης αυτής της διαδικασίας ε, και όταν θα φτάσουμε στο σημείο των, ε, του, το, της εκταμίευσης των 44 δισεκατομμυρίων, τότε πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι το ποσό αυτό θα οδηγήσει στην αηφόρο ανάπτυξη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, αυτή η μείωση του χώρου για τους πολίτες. Ίσως ε, θα μπορούσαμε και εμείς το επιχειρηματικό μας περιβάλλον να το αλλάξουμε ώστε να μπορεί να συμπεριλάβει περισσότερο χώρο για τους πολίτες και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό και η ΕΤΕ πρέπει να το λάβει υπόψη πολύ σοβαρά. Είναι γεγονός αν δεν υπάρχει χώρος ε, για την κοινωνία των πολιτών, δεν υπάρχει λογοδοσία και δεν υπάρχει εγγύηση ότι τα χρήματα θα εξυπηρετήσουν το στόχο της ανάπτυξης. Ευχαριστώ πολύ. Ο Σάρλ Γκέρενς. Ναι, μόλις κάποιος είπε ότι το Συμβούλιο ήταν ο πρωταγωνιστής της ιδέας ότι πρέπει να καταπολεμήσουμε τη μετανάστευση γιατί για τις χώρες ε, υπάρχουν χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τις οποίες είναι πραγματικό πρόβλημα αυτό. Λοιπόν, αυτό πρέπει να τοποθετηθεί σε μία άλλη προοπτική από αυτήν που παρουσίασε η προοπτική η προσκεκλημένη μας από την Oxfam. Πρέπει λοιπόν να είναι κατάλληλος, αποτελεσματικός ε, και αηφόρος ο μηχανισμός που θα ε, επικρατήσει. Και αυτό το λέω για την καθαρά αναπτυξιακή πολιτική. Όσον αφορά τώρα την οικονομική ανάπτυξη, δεν σημαίνει οικονομική ανάπτυξη ότι μειώνονται οι φτωχοί. Αντιθέτω, πρέπει να δούμε τον αντίκτυπο αυτή τη δράση. Αν θέλουμε όλος ο κόσμος να υποφελείται από αυτήν την ανάπτυξη, ε, τότε υπάρχει ε, ένα ζήτημα δικαιοσύνης που έχει άμεση σχέση με την, ε, την κυβέρνηση και το πώς αυτή διαχειρίζεται την ανάπτυξη αυτή ώστε να είναι ίση πρόσβαση όλων. Αυτό θα έδινε τη δυνατότητα σε όλους να υποφεληθούν από την ανάπτυξη Πρέπει να διαρθρωθούν ε, οι μηχανισμοί ε, που δημιουργούν νέες, ε, νέο πλούτο κατά αυτόν τον τρόπο. Θέλουμε να υπάρξουν, υπάρχει μια υποχρέωση για τα αποτέλεσμα, αλλά υπάρχει ελευθερία για τα μέσα. Αυτό που θα ήθελα να πω και το είπα και προηγουμένως, εγώ είμαι καταρχήν σύμφωνος αρκεί να ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις που έγιναν εδώ. Πρόκειται για μια αρκετά δύσκολη κατάσταση, είναι σπαζοκεφαλιά. Ε, όταν θα αρχίσουμε λοιπόν να δημιουργούμε μηχανισμούς πλούτου δεν σημαίνει ότι παντού θα είμαστε επιτυχείς. Ε, οι μόνες πτυχές ε, που θα ε, τονιστούν θα είναι οι αποτυχίες. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια ολόκληρη παιδαγωγική γιατί οι δημαγωγοί θα σύρουν το χορό όσον αφορά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων. Εκείνοι κάθε φορά θα λένε ότι θα υπάρξει ένα πρόβλημα που κάποιο θα βάλει το χέρι στο σάκο με τα χρήματα. Αυτό θα υπάρξει οπωσδήποτε. Κάποια στιγμή πάντοτε θα, ε, θα, θα, θα, θα υπάρξει ε, ε, κάποιος που δεν θα είναι τίμιος. Αλλά αυτό που πρέπει εμείς να εξηγήσουμε στην κοινή γνώμη είναι ότι το γεγονός ότι μια αποτυχία ε, δημοσιεύεται είναι η αποκάλυψη ενός συστήματος ελέγχου. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να υπάρξει πραγματικά προσπάθεια ε, εκπαίδευσης ως προς αυτό και πρέπει και να σχετικοποιήσουμε 1,5 δις θα ξοδέψουμε σε 65 ε, δις που ε, χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη, μπορούμε να αναλάβουμε τον ε, κίνδυνο μία τέτοια δαπάνη. Ε, αν υπάρχει ένας αντίκτυπος μόχλευσης από τις επενδύσεις από αυτό το 1,5 δις και ότι αυτό θα είναι ορατό στι ενδιαφερόμενε χώρες. Είναι πάντως παζοκεφαλιά αυτό, γιατί... Οι χώρες που το έχουν ανάγκη αυτό είναι οι χώρες με τη φτωχότερη διακυβέρνηση και θα ήθελα να σας ρωτήσω Πώ θα το αντιμετωπίσετε αυτό το θέμα. Πολύ διαφθαρμένε χώρε, ε, στις οποίες ε, κανονικά μέσω ε, ε του κανονικού προπολογισμού δεν δίνει χρήματα Ευρωπαϊκή Ένωση, μόνο μέσω προγραμμάτων. Πολύ έμεσα δηλαδή. Πώ θα οργανωθείτε λοιπόν στι χώρε αυτέ που είναι πολύ διαφθαρμένες, ε, ώστε να εξασφαλίσετε ότι ο κόσμο δεν θα μεταναστεύσει, συμφωνώ με την κυρία Χάουτελα και με την Όξφαμ ω προς αυτό, αλλά να υπάρχουν προοπτικές για τον κόσμο επιτόπου. Πώς κάνετε αυτό, πώς θα το καταφέρετε αυτό, είναι ένα κεντρικό ζήτημα το οποίο κατά τη γνώμη μου δεν το έχουμε καλύψει. Ναι, θέλω να δω πραγματικά γιατί η αναλογία του προπολογισμού μιλούμε. Κάποια στιγμή είναι σαν να λέμε ότι είναι ολόκληρο ο προπολογισμό ανάπτυξη. Όχι. Είναι μια πτυχή του συνολικότερου προπολογισμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τι Ανάπτυξη. Και συμφωνώ απολύτω ότι το να δώσουμε ελπίδα στη νέα γενιά της Αφρικής πρέπει να το κάνουμε, πρέπει ε, όπως και να το ονομάσουμε καταπολέμηση της φτώχειας, όπως θέλουμε να το πούμε, πρέπει να τους δώσουμε την ελπίδα ότι η ζωή τους θα γίνει καλύτερη. Και αυτό γιατί αυτός είναι ο απότερος στόχος ε, της αναπτυξιακής πολιτικής που θέλουμε να ε, επιτύχουμε. Φραντσέσκο Ραϊμόντι από την ΕΙΕΔ. Σύντομα όμως, γιατί έχουμε τον Επίτροπο που τον περιμένουμε σε πέντε λεπτά. Δεν θέλετε να πείτε κάτι. Α, εντάξει. Δεν είστε υποχρεωμένοι. Να δώσω τώρα το λόγο στους προσκεκλημένους για να μας απαντήσουν σε αυτά που άκουσαν. Δεν υπήρξαν συγκεκριμένες ερωτήσεις, αλλά θα δώσω και τη δυνατότητα στην Επιτροπή να απαντήσει. Ναι, ορισμένα πράγματα θα ήθελα να τα θέσω σε ένα πλαίσιο, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αφού μιλάμε για το εξωτερικό παιδίτικό σχέδιο κλπ. Υπάρχει μια ολοκλήρη συζήτηση ε, στον ΟΑΣΕ και στην αναπτυξιακό κομμάτι του ΟΑΣΕ ε, με πολύ σημαντικέ συνέπειε στην όλη διαδικασία. Ο συγχρονισμό των μέσων για τον ιδιωτικό τομέα ε, κυρίως η ευελιξία των κριτηρίων ε, για την επιλεξιμότητα των αναπτυξιακών προγραμμάτων ε, και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί αυτή η συζήτηση μπορεί να έχει αντίκτυπο και σε αυτό το ζήτημα που συζητούμε. Πώς λοιπόν η αναπτυξιακή βοήθεια που λογικά πρέπει να καταπολεμά τη φτώχεια και να βοηθά στην αξιοπρέπεια ε, πώς μπορεί λοιπόν να είναι ευέλικτη όλη αυτή η διαδικασία για να χρησιμοποιείται στον ιδιωτικό τομέα με την πρόθεση δημιουργίας ανάπτυξης και με την προϋπόθεση καταπολέμησης στόχες. Υπάρχει πάντα ένα κίνδυνο. και ο στόχος, η συζήτηση αυτή είναι πολύ σημαντική, όχι μόνο για το συγκεκριμένο στόχο, αλλά και για την ολόκληρη συζήτηση γύρω από την ανάπτυξη, στην οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πολύ δραστήρια. Ε, κοιτάξτε, εγώ δεν θα πρέπει, ξέρω ότι δεν πρέπει να αρνήσει όταν σου δίνουν το λόγο. Απλώ θα ήθελα απλώ να σα ευχαριστήσω για τη συζήτηση αυτή. Ελπίζω ότι δεν είναι η τελευταία φορά που έρχομαι και αναμένω αγωνίω μία ακόμη ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας ε, και άλλες πρωτοβουλίες, ε, μεταξύ των οποίων ε, την πρωτοβουλία αντοχής, όπως επίσης και την πρωτοβουλία επένδυσης ναι, βεβαίω, λέει η Πρόεδρο, ε, ενδεχομένω ε, να προσκαλέσουμε του συναδέλφου για το θέμα αυτό που ενδιαφέρει και πάρα πολύ και την κυρία Χάουταλα. Δίνω το λόγο σε εσά τώρα. Ναι, δύο ακόμη σημεία ε, θα ήθελα να τονίσω. Η προσθετικότητα, το είπα άλλωστε και στην, στα εισαγωγικά μου σχόλια, υπάρχει μια αξιολόγηση αυτού του blending, αυτή της συγχώνευσης που έδειξε πολύ θετικά αποτελέσματα. Θα ολοκληρωθεί και θα δημοσιευθεί σε, μια, σε ένα μήνα. Η λογοδοσία είναι ένα κεντρικό ε, σημείο της πρωτοβουλίας ε, για το blending. Από τα 2,7 δις ε, που επενδύσαμε στο blending σε σχέση με 278 ε, projects 250 ε, δισεκατομμυρίων. Θα έλεγα λοιπόν ότι ένα ευρώ που φεύγει από την ανάπτυξη είναι ένα ευρώ που προσελκύει πιο πολλά, ε, πιο πολλά χρήματα για την ανάπτυξη. Έτσι πρέπει να το βλέπουμε και για την κοινωνία των πολιτών νομίζω τα είπα όλα στην αρχή, δεν έχω τίποτε να προσθέσω και το ίδιο, το ίδιο ισχύει για την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια, δεν έχω τίποτε άλλο να πω, τα είπα στα εισαγωγικά μου σχόλια όλα. Ευχαριστώ ε, να ξανασυζητήσουμε μετά από την ε, τεχνική ενημέρωση και πιστεύω ότι όλα τα τεχνικά και τα οικονομικά ζητήματα θα έχουν αποσαφινιστεί και θα μπορέσουμε να ε, ολοκληρώσουμε ομαλά τις διαπραγματεύσεις. Καταρίνα, ναι ευχαριστώ πολύ σύντομα. Νομίζω κυρία Πρόεδρε, το είπατε κι εσείς πάρα πολύ σωστά και νομίζω ότι αυτό είναι το μήνυμα όταν μιλούμε για την υγεία, την εκπαίδευση, την κοινωνία των πολιτών, ε, μιλάμε για ένα τμήμα της ε, βοήθειάς μας, της συνολικής Νομίζω ότι το ιστορικό που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την υποστήριξη της κοινωνίας των πολιτών είναι πολύ σημαντικό, αλλά αυτό δεν είναι τμήμα διοχέτευσης όλων αυτών των μέσων, γιατί τα μέσα αυτά δεν αφορούν αυτό, μιλούμε για την ουσία. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ που το τονίσατε αυτό κυρία Πρόεδρε και κάτι ακόμη που θα ήθελα να πω ε, σε σχέση με τα σχόλια της Oxfam Θα δείτε νομίζω μία εξέλιξη μεταξύ της ε, ανακοίνωσης του Ιουνίου και του Σεπτεμβρίου. Ε, ακούσαμε δηλαδή πράγματι ε, και μας απασχόλησαν η ποικιλία των απόψεων των εμπλεκομένων φορέων, αλλά όσον αφορά το blending με τον ιδιωτικό τομέα, ας μην τα μπερδεύουμε. Αυτό αφορά τους διεθνούς αναπτυξιακούς εταίρους μας. Δεν έχουμε blending με τον ιδιωτικό τομέα ακόμη. Οπότε δεν ε, ε, προσπαθούμε να κάνουμε καμία παράκαμψη, προσπαθούμε να κάνουμε ένα blending σε ένα μικρότερο μέσο, γιατί ελπίζουμε έτσι να προσελκύσουμε τον ιδιωτικό τομέα. Συμφωνώ λοιπόν ε, μαζί σας ότι αυτό το blending με τον ιδιωτικό τομέα μπορεί να είναι κάποιο είδους παράκαμψη, αλλά είναι σημαντικό να γνωρίζει η Επιτροπή σας ε, ότι μπορεί να συμφωνούμε με κάποια από αυτά που ε, μας είπατε όταν θα έχουμε τα στοιχεία μπροστά μας και θα υπάρχει ένας ε, ένα συνδυασμός, ένα, ένα blending με συγκεκριμένα πρακτικά αποτελέσματα πόσο τυκοποιημένα και ένα νέο ε, στοιχείο, ένα νέο μέσο που προσπαθούμε να συμπεριλάβουμε στον ιδιωτικό τομέα, τότε θα είναι πιο σαφή τα πράγματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ όλους που προσήλθατε εδώ. Είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα και είδατε πόσο ενδιαφέρει τους ε, συναδέλφους. Είναι καλό που έγινε η συζήτηση τώρα, στην αρχή της διαδικασίας, ώστε να μπορούμε να έχουμε το σωστό σωστό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ.

Να καθίσουμε για να κάνουμε για να συζητήσουμε το τελευταίο θέμα της σημερινής μας συνεδρίασης. Είναι όμως πολύ σημαντικό το θέμα αυτό. Γιατί είναι μαζί μας ο Χρήστος Τηλιανίδης, που είναι όχι μόνο επίτροπος, αλλά και φίλος της επιτροπής μας. Ανέλαβε το χαρτοφυλάκιο του όταν σε μια περίοδο που η ανθρωπιστική βοήθεια ε, βρέθηκε στην εμπροστοφυλακή της παγκόσμιας ε, ατζέντα. Βρεθήκαμε πρόσφατα και στο Στρασβούργο όπου συζητήσαμε το ζήτημα της, ε, των ανθρωπιστικών κρίσεων. Έχουμε μπροστά μας το ενδεχόμενο να αντιμετωπίσουμε νέες ανθρωπιστικές κρίσεις στη Μοσούλη, στη Ράκα, τον ε, τυφώνα Μάθιου πρόσφατα στην ε, Καραϊβική. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε σήμερα λοιπόν είναι να συζητήσουμε τα σχέδια για του χρόνου, για το 2017, τις προτεραιότητες της ανθρωπιστικής βοήθειας και αυτά θέλουμε να συζητήσουμε μαζί σας. Παρ' όλα αυτά να σημειώσω την ε, πολύ βαθιά εκτίμηση Τη Επιτροπής μας για το έργο που επιτελείτε εσείς και το επιτελείο σα σε πολύ πολύ δύσκολες συνθήκες. Κύριε Επίτροπε, έχετε τον λόγο. Γνωρίζετε λοιπόν ότι είμαστε όλοι στην ίδια κατάσταση, αντιμετωπίζουμε τα ίδια προβλήματα και για μας, για όλους μας, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει συνεργασία μεταξύ ημών και ημών και εδώ στις Βρυξέλλες, αλλά ε, ιδίως και στους ε, στις περιοχές όπου μένονται τα προβλήματα. Αγαπητοί συνάδελφοι, λοιπόν, χαίρομαι κάθε φορά που βρίσκομαι εδώ στην οικογένειά μου, όπως έχουμε πει και άλλες φορές για την σχέση που έχω μαζί σας. Χαίρομαι πολύ που σας βλέπω και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Δυστυχώς, οι ανθρωπιστικές κρίσεις ε, βρίσκονται, ε, διάφορες ανθρωπιστικές κρίσεις βρίσκονται σε εξέλιξη. Οι ανάγκες αυξάνονται στη Μέση Ανατολή, στην Αφρική και φυσικά στην Κεντρική Αμερική. Αλλά ας μην ξεχνάμε βεβαίως και την ε, προσφυγική κρίση εντός της Ευρώπης. Ταυτόχρονα πρέπει να ομολογήσουμε ότι το ευρωπαϊκό εγχείρημα, η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει πρωτοφανείς προκλήσεις. και είναι και αυτό μια πολιτική, ένα πολιτικό καθήκον που έχουμε είτε ως επίτροποι είτε ως ευρωβουλευτές, ως ηγέτες αυτών των θεσμικών οργάνων. Παρόλα αυτά, μέσω της ανθρωπιστικής βοήθειας επιτόπου αποδεικνύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει ένας από τους πυλώνες της παγκόσμιας δράσης. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να μιλήσω για αυτή την πρωτοφανή προσφυγική κρίση που βιώνουμε. Τον Μάρτιο παρουσίασα στην Επιτροπή σας αυτό το νέο εργαλείο για την υποστήριξη έκτακτης ανάγκης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ιδίως την δική σας Επιτροπή για την υποστήριξή σας και για, το, για τα κονδύλια που κατανεμήθηκαν. Μέχρι στιγμής περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ έχουν διατεθεί μέσω των εταίρων μας στην ανθρωπιστική βοήθεια για τα ε, project μας στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα υπάρχουν πάνω από 60.000 πρόσφυγες. Σε αυτό το στάδιο λοιπόν οι απαντήσεις που δίνουμε επικεντρώνονται σε τέσσερις προτεραιότητες. Πρώτον, την προετοιμασία των υπαρχόντων καταβλισμών για τους κρύους μήνες του χειμώνα. Δεύτερον, την παροχή βοήθειας μέσω μετρητών και βάουτσερ, και αυτό είναι σημαντικό και θα σας εξηγήσω γιατί. Τρίτον, την παροχή εκπαίδευσης για τα παιδιά σε αυτές τις πολύ δύσκολες συνθήκες. Και τέταρτον, την παροχή φροντίδας στους ασυνόδευτού ανήλικους που είναι η πλέον ευάλωτη πληθυσμιακή ομάδα και ταυτόχρονα η πιο τραγική πλευρά αυτής της πρωτοφανής κρίσης. Έπειτα από πολλά εμπόδια και πολλές προσπάθειες που καταβλήθηκαν με τις, σε συνεργασία με τις ελληνικές αρχές, τα αποτελέσματα είναι ήδη απτά. Συνεχίζεται η προετοιμασία για τον χειμώνα, τον καταβλισμό των προσφύγων και ταυτόχρονα διανέμονται ήδη για τον χειμώνα από τους εταίρους μας, τόσο στην υπηρετική χώρα όσο και στα νησιά της Ελλάδας. Ταυτόχρονα προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε ότι 9.000 παιδιά θα έχουν δυνατότητα μετακίνησης από και προς τα δημόσια σχολεία, ότι θα έχουν βασικά σχολικά είδη για να μπορέσουν να μάθουν να διαβάζουν και να γράφουν. Συνεργαζόμαστε με τις τοπικές αρχές και άλλους εταίρους προκειμένου να αυξήσουμε τον, ε, τους χώρους φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων. Ενισχύουμε τις δομές φροντίδας και ιατρικής περίθαλψης, ψυχολογικής υποστήριξης αλλά και ψυχαγωγίας για τους ε, ασυνόδευτους ανήλικους. Ταυτόχρονα έχουμε μέσω του μηχανισμού πολιτικής προστασίας διανύμει χιλιάδες είδη ανακούφισης σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στις υπόλοιπες χώρες της περιοχές. Και γι' αυτό θα ήθελα να σας υποδεχθώ τις επόμενες εβδομάδες σε αυτό το συντονιστικό κέντρο ε, απάντησης και διαχείρισης κρίσεων που ε, για να σας δείξω με ποιον τρόπο θα καταφέρουμε να καταβάλουμε αποτελεσματικές προσπάθειες για την επίλυση των προβλημάτων. Να περάσω τώρα στην Τουρκία. Η διευκόλυνση για τους πρόσφυγες βρίσκεται σε λειτουργικό στάδιο πλέον και αποφέρει θετικά αποτελέσματα παρά τα πολιτικά εμπόδια που έχουμε αντιμετωπίσει. Ε, ε, ε, από τις αρχές του 2016 πάνω από 1,25 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν δοθεί με τη μορφή συμβάσεων. 512 εκατομμύρια έχουν διατεθεί άμεσα για την ανθρωπιστική βοήθεια. Και στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας η διευκόλυνση για την Τουρκία έχει χαράξει το δρόμο για ένα ριζοσπαστικό ε, δίκτυο ασφαλείας κοινωνικών κρίσεων, που είναι το μεγαλύτερο ανθρωπιστικό πρόγραμμα που χρησιμοποιεί άμεσα τις μεταφορές μετρητών μέχρι σήμερα. Κοιτάξτε τι καταφέραμε να κάνουμε με τα 348 εκατομμύρια ευρώ που διατέθηκαν μέσω του ESSN. Σε συνεργασία με το Παγκόσμιο Επιστημιστικό Πρόγραμμα, τον, ε, την ε, τουρκική Ερυθρά ημισέλινο και βεβαίως τις τουρκικές αρχές, βοηθήσαμε ένα εκατομμύριο από τους πλέον ευάλωτους πρόσφυγες στην Τουρκία. Η μεγαλύτερη πλειονότητα αυτών ζει εκτός καταβλισμών. Και μέσω αυτού του Cash and Vouch ε, Scheme καταφέραμε να δώσουμε ψωμί σε αυτούς τους ανθρώπους. Μια στέγη πάνω από τα, κεφάλια, από τα κεφάλια τους και οι άνθρωποι αυτοί χάρη στις προσπάθειές μας, μπορούν να στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Με μεγάλη περηφάνεια μπορώ να προσθέσω ότι το ESSN είναι και εξαιρετικά αποδοτικό από οικονομικής άποψης. 85% της συμβολής μας θα κατευθυνθεί απευθείας σε ευάλωτους πρόσφυγες και με αυτόν τον τρόπο υποστηρίζουμε και εξασφαλίζουμε, προστατεύουμε την, την αξιοπρέπεια των προσφύγων για ευνόητους λόγους. Ταυτόχρονα όμως προστατεύουμε και την τοπική οικονομία μέσω της βοήθειας προς τις μικρομεσές επιχειρήσεις. Αυτό είναι ένα στοιχείο που πραγματικά καθορίζει την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και είναι ένα στοιχείο, ένα μοντέλο που έχουμε αρχίσει σταδιακά να εφαρμόζουμε στην ε, Ελλάδα. Έχουμε συζητήσει και με πολίτες της Τουρκίας και έχουμε διαπιστώσει ότι αυτό το ε, σύστημα μετρητών και κουπονιών βοηθά τις τοπικές κοινωνίες, την κοινωνική ένταξη των προσφύγων και την εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ των προσφύγων και των τοπικών πληθυσμών. Αγαπητοί συνάδελφοι, η πρώτη μας προτεραιότητα όσον αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια είναι βεβαίως η κατάσταση στην Σύρια. Σχεδόν έξι χρόνια συγκρούσεων έχουν περάσει και παρόλα αυτά δυστυχώς δεν φαίνεται να υπάρχει διέξοδος. Πάνω από 13 εκατομμύρια άνθρωποι αντιμετωπίζουν επίγουσες ανάγκες στη Συρία και πάνω από 5 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν διαφύγει σε γειτονικές χώρες και στην Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος χρηματοδότης στην Συρία από, την, ε, από το ξέσπασμα της σύγκρουσης. Έχουμε κινητοποιήσει σχεδόν 9 δισεκατομμύρια ευρώ σε ανθρωπιστική βοήθεια και κονδύλια για την ανάπτυξη και την σταθεροποίηση. Ωστόσο, οι πραγματικά αποτρόπες επιθέσεις σε αμάχους, σε νοσοκομεία, σε σχολεία, ακόμη και σε κονβόι βοήθειας, βρίσκονται σε πλήρη παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Αυτά είναι όλα τα καταστροφικά αποτελέσματα της ε, επιδεινούμενης ανθρωπιστικής κατάστασης. Στο Ανατολικό Αλέπο 300.000 άνθρωποι έχουν αποκοπεί από κάθε είδους βοήθειας εδώ και δύο μήνες. Τα αποθέματα τροφίμων και φαρμάκων εξαντλούνται. Τον προηγούμενο μήνα η Φεντερίκα Μογκερίνη, είπατη εκπρόσωπος και αντιπρόεδρος της Κομισιόν, ξεκίνησε μια ανθρωπιστική πρωτοβουλία για το Χαλέπι σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη. Δύο ήταν οι βασικοί στόχοι που τέθηκαν. Πρώτον, το να παρασχεθεί βοήθεια στο Ανατολικό Χαλέπι και δεύτερον, να εκενωθούν και να διευκολυνθεί η εκένωση των τραυματιών και των πληγέντων. Η πρωτοβουλία έτυχε σημαντικής υποστήριξης και από το Κοινοβούλιο και γι' αυτό θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Παρ' όλα αυτά και δυστυχώς δεν έχουμε καταφέρει ακόμη να φτάσουμε σε όλους τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Συνεχίζουμε να ασκούμε πολιτικές πιέσεις και τονίζουμε και σε άλλους παγκόσμιους και περιφερειακούς παράγοντες και φορείς ότι ο σεβασμός του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου πρέπει να τεθεί σε πρώτη προτεραιότητα. Δυστυχώς όμως η κατάσταση επιδεινώνεται μέρα με τη μέρα. Επιμένουμε σε αυτήν την πρωτοβουλία. Εγώ και η Φεντερίκα συζητούμε με πάρα πολλούς τοπικούς φορείς με Ρώσους εταίρους τον κύριο Λαυρόφ. Κάποιες από τις ομάδες που δραστηριοποιούνται εντός της Συρίας με αξιωματούχους του καθεστώτος Ασάντ. Δυστυχώς όμως μέχρι στιγμής δεν έχουμε καταφέρει να ε, καταλήξουμε σε κάποιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Το δικό μας επιχείρημα είναι πολύ απλό. Η ανθρωπιστική βοήθεια χρειάζεται εγγυήσεις, όχι μόνο κατάπαυση πυρός. Χωρίς αυτές τις εγγυήσεις εμείς δεν είμαστε σε θέση να παράσχουμε την ανθρωπιστική μας βοήθεια. Να περάσω τώρα στο θέμα του Ιράκ όπου η κατάσταση έχει σημαντικότατες ανθρωπιστικές επιπτώσεις. Η συλλογική μας δράση εκεί πρέπει να συνεχιστεί. Πρώτα απ' όλα για να δοθεί μια απάντηση στις εξαιρετικά μεγάλες ανθρωπιστικές ανάγκες. Και δεύτερον, όπως και στη Συρία, δεν μπορεί να υπάρξει σταθερότητα στην περιοχή όσο βρίσκεται σε εξέλιξη η σύγκρουση. Με, δεδομένο, ε, με δεδομένες τις τελευταίες εξελίξεις στη Μοσούλη, θα ήθελα να επισημάνω ότι έχουμε προετοιμαστεί για ε, αυτήν την μέρα εδώ και μήνες. Εγώ συμμετείχα εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην συνδιάσκεψη που έγινε με θέμα το Ιράκ στην Ουάσιγκτον τον Ιούλιο έπειτα από πρόσκληση του Υπουργού Εξωτερικών, Κέρι. Έχω, συζητή, έχω επισκεφτεί τη χώρα τέσσερις φορές για να βεβαιωθώ ότι ήμασταν προετοιμασμένοι να ανταποκριθούμε στις ανάγκες που θα προέκυπταν στη Μοσούλη. Επισκέφτηκα τον καταβλισμό Μπάκα και τις προετοιμασίες που βρίσκονταν σε εξέλιξη εκεί. Πρέπει να σας πω ότι οι άνθρωποι μας ήταν προετοιμασμένοι προκειμένου να αντιμετωπίσουν μια ανθρωπιστική κρίση. Αλλά καθώς η κατάσταση βαίνει επιδεινούμενη, δυστυχώς πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι θα αντιμετωπίσουμε ανθρωπιστικές τραγωδίες. Μέχρι στιγμής τα πράγματα φαίνονται ότι βρίσκονται υπό έλεγχο. Αυτές είναι οι πληροφορίες που έχουμε από τους εταίρους μας που δρούν επιτόπου. Επιτρέψτε μου να πω και δύο λόγια για την Αφρική. Θα επισκεφθώ την Ουγκάντα την, ε, την Πέμπτη και την ε, Παρασκευή. για να σχηματίσω μια εικόνα για το πώς η χώρα αντιμετωπίζει την ε, μαζική εισρωή προσφύγων που προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο στο Νότιο Σουδάν. Μετά το ξέσπασμα των συγκρούσεων στο Νότιο Σουδάν το καλοκαίρι, 240.000 πρόσφυγες έχουν καταφτάσει στην Ουγκάντα από την 1η Ιουλίου. Αν συνεχιστεί η τάση αυτή ενδέχεται έως το τέλος της φετινής χρονιάς στην Ουγκάντα να ε, συγκεντρωθούν έως και ένα εκατομμύριο πρόσφυγες. Τα στοιχεία μιλούν από μόνα τους. Καμία χώρα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνη της τόσο μεγάλες προκλήσεις. Και παρόλα αυτά αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν πολλοί φορείς στην Αφρική, όπου η ευθραυστότητα και οι συγκρούσεις συνεχίζουν να πετούν εκατομμύρια ανθρώπους στο δρόμο και στην προσφυγιά. Δημιουργούνται ανθρωπιστικές κρίσεις που δεν την χάνουν ούτε καν της προσοχής των μέσων ενημέρωσης. Γι' αυτό και είναι σημαντικό να υψώσουμε τη φωνή μας και να συνεχίσουμε να επιδεικνύουμε την αλληλεγγύη μας με αυτούς τους πληθυσμούς που αντιμετωπίζουν τις πλέον πιεστικές ανάγκες. Αυτό νομίζω ότι είναι το σημαντικότερο στην περίπτωση της Ουγγάντα. Και γι' αυτό το λόγο θα επισκεφτώ και το Μαλάουι στα τέλη του Νοεμβρίου για να δω πώς μπορούμε να συνεχίσουμε την, ε, τις προσπάθειές μας για να δώσουμε βοήθεια ε, στους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν τις αρνητικές επιπτώσεις του φαινομένου ελληνίνιου. Για άλλη μια φορά θα ήθελα να τονίσω ότι δεν αρκεί από μόνη της η ανθρωπιστική βοήθεια. Πρέπει να, να δημιουργήσουμε ένα συνεχές προκειμένου η ανθρωπιστική βοήθεια να συμβάλλει στην ανθεκτικότητα, τη σταθεροποίηση και την ανάπτυξη. Αν δεν το καταφέρουμε αυτό, οι πρόσφυγες δεν θα είναι σε θέση ποτέ να επιστρέψουν στις αιστείες τους. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Γνωρίζω ότι πολλοί από εσά θεωρείται πάρα πολύ σημαντικό, σημαντική την τη σύνδεση αγωγής, αποκατάστασης και ανάπτυξης. Και δικαίως το κάνετε αυτό. Αντιμετωπίζουμε όλο και περισσότερες παρατεταμένες κρίσεις. Αυτό ήταν και ένα από τα ε, βασικά ε, μηνύματα που αποστήλαμε το τελευταίο διάστημα. Είμαστε αποφασισμένοι να εφαρμόσουμε τις 100 δεσμεύσεις μας στην πολιτική, επιχειρησιακά, αλλά και σε οικονομικά ζητήματα. Βεβαίως, ταυτόχρονα θα εξασφαλίσουμε το συντονισμό και με άλλους εμπλεκόμενους φορείς. Να ενώσουμε τις δυνάμεις μας σε αυτήν την διαδικασία που θα ακολουθήσει από εδώ και πέρα στο πλαίσιο του WHS σε μια σειρά δεσμεύσεις έχουμε ήδη αρχίσει να επιτυχάνουμε μετρήσιμα αποτελέσματα. Με τον συνάδελφο Επίτροπο Μίμητσα έχουμε προσδιορίσει πιλωτικές χώρες όπου θα επιχειρήσουμε να ενισχύσουμε τις συμπράξεις μας. Ένα εξαιρετικό παράδειγμα είναι η ανακοίνωση με τίτλο «Ζωές με αξιοπρέπεια» που εγκρίθηκε τον Απρίλιο. Βρισκόμαστε σε μια μεταβατική περίοδο με τελικό στόχο να, να, να καταφέρουμε να δώσουμε τη δυνατότητα στους εκτοπισμένους ανθρώπους να γίνουν περισσότερο αυτάρκης και να μπορέσουν να ζήσουν μια αξιοπρεπή ζωή. Γιατί πίσω από τους συγκλονιστικούς αριθμούς που βλέπουμε καθημερινά στις ειδήσει, να μην ξεχνούμε ότι κρύβονται άνθρωποι, άνθρωποι που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση απαντά ε, στην παγκόσμια κρίση εκτοπισμού. Πάνω από τα δύο τρίτα του ετήσιου προϋπολογισμού μας για την ανθρωπιστική βοήθεια αξιοποιείται για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων για πρόσφυγες, τους εσωτερικά εκτοπισμένους και τις ε, κοινότητες που τους έχουν υποδεχθεί. Σε, σε ευθυγράμμιση βεβαίως με τις ευρωπαϊκές αξίες και αρχές μας. Οι άνθρωποι αυτοί, δεν, δεν αποτελούν πηγή ανησυχία μόνο για εκείνους που παρέχουν ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά και για φορείς που ασχολούνται με την οικονομική ανάπτυξη. Αυτό ίσχυε πάντοτε, αλλά μέσω της έγκρισης, της υιοθέτησης αυτής της ολοκληρωμένης στρατηγικής καθιστούμε τις προσπάθειές μας πιο συστηματικές. Επίσης, σημαντική είναι η κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι, τα τρία εκατομμύρια Αφγανών προσφύγων στο Ιράν, που βρίσκονται εκεί εδώ και περισσότερες από τρεις δεκαετίες. Εγώ επισκέφθηκα τη χώρα πριν από δύο εβδομάδες και επισκέφθηκα τα προγράμματα που υλοποιούμε στη βάση με επικέντρωση στο θέμα της παιδείας. Και με αυτό θα ήθελα να περάσω στο επόμενο σημείο της ομιλίας μου. Οι πλέον ευάλωτοι άνθρωποι σε καιρούς κρίσης, το γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά, είναι τα παιδιά. Το να εξασφαλιστεί η ευημερία των παιδιών είναι κεφαλαιόδους σημασίας και γι' αυτόν τον λόγο η εκπαίδευση σε καιρούς έκτακτης ανάγκης εξακολουθεί να είναι η δική μου πρώτη προτεραιότητα. Ξέρω ότι είναι προτεραιότητα και για σας και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά για την υποστήριξή σας που μας ε, επέτρεψε να αυξήσουμε τον προϋπολογισμό πάνω από τέσσερις φορές με αποτέλεσμα να καταφέρουμε να φτάσουμε και να βοηθήσουμε 2,3 εκατομμύρια παιδιά σε 44 χώρες. Σε αυτόν τον τομέα η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πραγματικά επικεφαλής, πρωτοπόρος με το παράδειγμά της και έχουμε κάθε πρόθεση να συνεχίσουμε ακατάπαυστα τις προσπάθειές μας και σε αυτόν τον τομέα. Έχουμε μια νέα αξιολόγηση προκειμένου να καθοδηγούνται οι δικές μας προτεραιότητες, μια αξιολόγηση για την προστασία των παιδιών και των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και το βασικό συμπέρασμα είναι ότι έχουμε ήδη επιτύχει σημαντικότατα αποτελέσματα, ιδίω όσον αφορά τους πρόσφυγες και τους εσωτερικά εκτοπισμένους ανθρώπους. Ταυτόχρονα όμως υπάρχουν και περιθώρια βελτίωσης και γι' αυτόν τον λόγο του επόμενου μήνε θα εξετάσουμε τα επόμενα βήματα που θα αναλάβουμε όσον αφορά την πολιτική μας αλλά και τη στρατηγική μας προσέγγιση αλλά και για τις συμπράξεις και τις συνέργειες που μπορούμε να αναλάβουμε με τους συναδέλφους μας που ε, εργάζονται στον τομέα της οικονομικής ανάπτυξης. Όπως ξέρετε, το θέμα της ανθεκτικότητας είναι κάτι που μας απασχολεί. Ελέγχουμε την κατάσταση εκ του σύνεγγης με αυτό το πρόγραμμα δράσης Sendai, το οποίο εκπονήσαμε φέτος τον ε, Ιούνιο. Έχει μεγάλη σημασία να αναπτύξουμε την ανθεκτικότητά μας για να καταφέρουμε περισσότερα με λιγότερα μέσα. Αυτό είναι και το μεγάλο μας στίχημα. Θα ήθελα τέλος να αναφερθώ σε ένα νέο μέσο που ε, προέβαλε ο πρόεδρος ε, Γιούνκερ κατά την ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης. Πρόκειται για ένα εθελοντικό σώμα βοηθείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε μέσω ενός ε, σώματος εθελοντισμού. Η Επιτροπή θα σας υποβάλει περαιτέρω λεπτομέρειες τον Δεκέμβριο. Πιστεύω ότι έτσι θα βελτιώσουμε τη λειτουργία μας και θα δώσουμε νέες ευκαιρίες στη νέα γενιά. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να ολοκληρώσω με ένα προσωπικό σχόλιο. Με τιμά η υποστήριξή σας εδώ και δύο χρόνια κατά την φιτία μου. Είμαι ευγνώμων γιατί μπορώ να βασιστώ στη συνεργασία σας, το, τα δικά σας σχόλια, ανησυχίες, υποδείξεις και ιδέες. Είτε από την Επιτροπή ΔΕΒΕ, είτε και διμερός. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι σίγουρος ότι μπορούμε να συνεχίσουμε αυτή την πολύ επικοδομητική συνεργασία μέσα στα πλαίσια των κοινών μας υποχρεώσεων και καθηκόντων και νομίζω ότι υπάρχει περιθώριο να βελτιώσουμε και να βελτιωθούμε, όπως ε, πάντα. Περιμένω τα σχόλιά σας και τις ε, επικρίσεις σας εκεί όπου χρειάζεται. Σας ευχαριστώ. Um, thank you, Commissioner. And thanks Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή σας την εισήγηση και απολογισμό. Βλέπουμε ότι υπό δύσκολες συνθήκες η επιτόπια, η εργασία είναι ύψης της ε, σημασίας. Έχουμε και εκπροσώπους από ΜΚΟ που εργάζονται υπό σκληρές συνθήκες. Ο κύριος Ενρίκε Γκερέος Σαλόμ. Είναι 6 και 5. Πρέπει να ολοκληρώσουμε στις 6.30. Ο και θα λάβει καταρχήν το λόγο. Θα ήθελα να κάνω ορισμένα σχόλια και ερωτήσεις. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο, τον κύριο Στυλιανίδη, γιατί προσέρχεται συχνά στην Επιτροπή μας και ε, συναντάτε μαζί μας ε, επίσημα ή ατύπως, όποτε χρειάζεται. Το θέμα της ανθρωπιστικής βοήθειας ε, είναι πιο ειρηνικό σε σχέση με την ανάπτυξη, όπου έχουμε πολλές συγκρούσεις. Κάθε χρόνο αυξάνεται ο αριθμός των ανθρώπων που χρήζουν ανθρωπιστικής βοήθειας και τα επόμενα χρόνια θα διονγκώνεται ο αριθμός τους. Πρέπει να συγχαρούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί πέρσι αύξησε κατά 35% την ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για την ε, υποστήριξή της. Ο Επίτροπος μίλησε για την ανάγκη το να είμαστε ένας παγκόσμιος παίκτη στη χορήγηση ανθρωπιστικής βοήθειας και μας απασχολούν οι ανθρωπιστικές κρίσεις ε, πολύ κοντά μας, ε, στη γειτονιά μας θα μπορούσα να πω. Μιλώ για το Ιράκ και τη Συρία. Υπάρχουν όμως και άλλες συγκρούσεις ανά τον κόσμο. Αναφερθήκατε στην Ουγκάντα Αύριο προβλέπεται μία συγκεκριμένη ε, δράση του Κοινοβουλίου για το ε, τρίγωνο της, ε, των Ονδουρών, του Ισημερινού και της Γουατεμάλας. Θα πρέπει λοιπόν να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να αντιμετωπίσουμε τις κρίσεις όπου και να υπάρχουν. Μιλήσαμε και για την κρίση του έμπολα, της ΑΙΤΙΣ και του Ισημερινού. Θα ήθελα να τονίσω ότι στην Επιτροπή αυτή ανησυχούμε ιδιαίτερα ως προς τους ε, συνοριακούς ελέγχους και τη διανομή της ανθρωπιστικής βοήθειας. Πριν υποβάλω τις ερωτήσεις, θα ήθελα να πω ότι έχω μπροστά μου μία έκθεση του Norwegian Refugee Council που μιλά για προετοιμασία για τις ε, ε, κρίσεις πριν επέλθουν. Μιλάμε και για την προετοιμασία αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, αλλά και την επίλυση συγκρούσεων. Δεν ξέρω κατά πόσο η Γενική Διευθυνσή ΕΚΟ θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις ξεχασμένες κρίσεις και θα προωθήσει την ανθρωπιστική βοήθεια μέσα στα πλαίσια του Enhanced Response Capacity. Έπειτα, Κατά δεύτερον, θα ήθελα να ρωτήσω κατά πόσο θα υπάρχει μια υψηλότερη προβλεψιμότητα της ανθρωπιστικής βοήθειας για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε άμεσα τη στιγμή που ενσκύπτουν ανθρωπιστικές κρίσεις. Επίσης, έχει σημασία να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια και προβλεψιμότητα των, ε, της βοήθειας εκεί όπου χρειάζεται, με βάση τα μέσα που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχω πέντε ομιλητές, δύο λεπτά ο καθένας. Σας διαβάζω. Πεθέρα, Ignacio Maria Norbert Neuser and Αυτοί είναι οι ομιλητές. Δύο λεπτά για τον καθένα για να μπορέσει να απαντήσει ο Επίτροπος. Η Μπεατρίφ. ευχαριστώ. Καταρχήν θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον Επίτροπο Στυλιανίδη γιατί είναι πάντα διαθέσιμος και γιατί πάντα προσπαθεί να ασχοληθεί εις βάθος με το ζήτημα και με επιμέρους ζητήματα που πολλές φορές είναι ε, έστω και λίγο εκτός των αρμοδιοτήτων του. Με βάση αυτά που είπε και ο και Γκερέρο, πέρα από την λυπηρή κατάσταση που μας παρουσίασε και με την ανθρωπιστική κρίση που βρίσκεται πολύ κοντά μας, θα θέλαμε να ασχοληθούμε και με την Κεντρική Αμερική, όπως υπενθύμησε ο Ενρίκε. Ε, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω και την Βενεζουέλα. Η Βενεζουέλα ζει μια μεγάλη ανθρωπιστική κρίση, δεν υπάρχουν φάρμακα, τρόφιμα, δεν υπάρχουν ε, πηγές ενέργειας και όλα επιδεινώνονται. Νομίζω ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να μιλούμε για τη Βενεζουέλα και να συνεισφέρουμε εκεί όπου μπορούμε γιατί μπορεί να μην μας το ζητούν επίσημα, αλλά θα πρέπει να το έχουμε κατά νου. Επίσης ε, και κάτι άλλο, στην Ελλάδα που βρέθηκα την προηγούμενη εβδομάδα, είδα την κατάσταση στα κέντρα υποδοχής ε, και στο ελληνικό και στο Σκαραμαγκά. Γνωρίζω τα προβλήματα που υπάρχουν και αντιμετωπίζει η ελληνική κυβέρνηση, αλλά αυτό που με ενδιαφέρει ιδιαίτερα είναι οι μη συνοδευόμενοι ανήλικες. Πέρα από το γεγονός ότι δεν μπορεί να υπάρξει παραδειγματική υποδοχή αυτών των ανηλίκων πάντα, θα ήθελα να λάβω υπόψη να μου πείτε μάλλον γιατί δεν αντιμετωπίζει ε, την κατάσταση τόσων ανηλίκων γιατί ε, μόνο υπάρχουν 1.700 ανήλικες που περιμένουν μια διαδικασία υποδοχής και έχουν τύχει υποδοχής μόνο 36 από όσο μου ελέγχθη. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε κατά πόσο μπορεί να ανταποκριθεί η Ελλάδα σε αυτή την κατάσταση που αφορά τους ε, ανήλικες. Γιατί δεν μιλάμε για αλληλεγγύη, μιλάμε για νομική υποχρέωση. Πολύ καλή ερώτησή σας. Ο Ιγνάσιο Κοράου και μετά η Μαρία. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας κύριε Επίτροπε. Σε δύο λεπτά μερικές ερωτήσεις θα ήθελα να θέσω. Το πρώτο ερώτημα είναι ότι είναι ευρέως αναγνωρισμένο ότι συχνά συγκρούσεις που έχουν ε, να κάνουν με ε, περιβαροντικούς και φυσικούς ε, λόγους, όπως για παράδειγμα στον Μπαγκλαντές, ε, όπου υπήρχαν πάρα πολλά προβλήματα τα οποία εκμεταλλεύτηκαν οι στρατιωτικές δυνάμεις της Ονδούρας, που είχε, που είχε σημαντικό αποτέλεσμα στον τοπικό πληθυσμό. Η Κολομβία έχει... βρίσκεται σε παρόμοια κατάσταση, όπου παραστρατιωτικές οργανώσεις έχουν αναλάβει τα ε, η ε, και υπάρχουν τώρα απειλές προς τους ντόπιου να φύγουν από την ε, Κολομβία. Πάρα πολλοί άνθρωποι λοιπόν υποφέρουν επειδή αποτελούν εμπόδιο στην επιδίωξη οικονομικών καθαρά Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Πώς ακριβώς προσπαθείτε να λύσετε τέτοια προβλήματα και να τα αποφύγετε ε, θα μπορέσει η παρέμβασή σας να είναι ορατή. Ε, όσον αφορά τον, Ιταλ... τον σεισμό στην Ιταλία τώρα, η Ιταλία δεν ζήτησε βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση παρά το γεγονός ότι εσείς το είπατε στην τελευταία σας δήλωση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την πρόθεση και είναι έτοιμη να βοηθήσει την Ιταλία ε, να αντιμετωπίσει τις συνέπειες του σεισμού. Ε, έχετε, ποια είναι η άποψή σας σε σχέση με το γεγονός ότι η Ιταλία δεν ζήτησε βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε που βρίσκεστε εδώ σήμερα και σας ευχαριστώ και για τις ε, δραστηριότητες σας και για το έργο σας για τα παιδιά. Θέλω να επικεντρωθώ σε ένα ε, σημείο. Είπατε ότι θα πάτε στο Μαλάουι για να παρακολουθήσετε και να αξιολογήσετε τις επιπτώσεις του Ελληνίνιου Εγώ βρέθηκα στη χώρα το καλοκαίρι και είναι ένα πραγματικά κλασικό παράδειγμα. Πρώτα υπήρξαν πλημμύρες, εκτοπίστηκαν οι χώρες αυτές και οι οικογένειες αυτές ε, που ζούσαν στις περιοχές αυτές και τώρα αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της ξηρασίας. Έχω την αίσθηση λοιπόν ότι βρισκόμαστε διαρκώς σε μια διαδικασία να κυνηγούμε την, την ουρά μας στην ουσία. Ε, και αυτό σχετίζεται με το γεγονός ότι δεν έχει ακόμη οικοδομηθεί μια ανθεκτική γεωργία. Θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα αν μιλούσαμε απλώς για, ε, την, ε, για πολέμους. Εδώ όμως, σε αυτό το, σε αυτό το τομέα, βρίσκω ότι βρισκόμαστε, είμαστε ουραγοί όσον αφορά τις σύγχρονες μεθόδους γεωργίας. Και ε, είναι ιδιαίτερα εμφανές αυτό το πρόβλημα στην στην Αφρική. Είπατε για την μείωση των κινδύνων από τις φυσικές καταστροφές. Πώς μπορούμε να ασκήσουμε ακόμη μεγαλύτερες πιέσεις προκειμένου να περάσουμε σε συστήματα ανθεκτικότερα από αυτά που έχουμε σήμερα. Επειδή λοιπόν δεν έχουμε πολύ χρόνο, θα ήθελα για άλλη μια φορά να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς εσάς για, το πραγματικά ε, εξαιρετικό έργο σας. Ο κύριος Νόιζερ. Κύριε Επίτροπε, είναι πραγματικά πολύ θετικό το γεγονός ότι βρίσκεστε σήμερα εδώ μαζί μας. Δύο συγκεκριμένα ερωτήματα έχω να σας θέσω. Κατά 35% αυξήθηκαν τα κονδύλια. Ερώτημα. Ήταν αρκετά προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι κρίσεις που αντιμετωπίζουμε. Δεύτερο ερώτημα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπόρεσε να βοηθήσει την ύπατη αρμοστία ε, ε, και τη UNICEF για την αντιμετώπιση των κρίσεων ή εκκρεμούν ακόμη ε, πληρωμές από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βρέθηκα την προηγούμενη εβδομάδα στο Λίβανο. Είναι πραγματικά κρίσιμη η εκρεμουν ακομη ε πληρωμες απο την πλευρα της ευρωπαικης ενωσης βρεθηκα την προηγουμενη εβδομαδα στο λιβανο ειναι πραγματικα κρισιμη η κατασταση 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες έχουν συγκεντρωθεί στη χώρα, 400.000 παιδιά σε ηλικία σχολική βρίσκονται εκεί. Οι πιέσεις που ασκούνται στα σχολεία είναι τεράστιες. Τα σχολεία δεν λειτουργούν με βάρδιες πλέον. Παρόλα αυτά, το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τον, ε, τους πρόσφυγες αλλά και τον λιβανέζικο πληθυσμό. Γι' αυτό και αξίζει η χώρα της δικής μας υποστήριξης. Και χαίρομαι που είπατε ότι πρέπει να μιλήσουμε και για την βελτίωση της ε, κατάστασης γύρω από την υγιεινή αλλά και όσον αφορά την αποκομιδή των σκουπιδιών γιατί 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι είναι εύλογο ότι δημιουργούν τεράστιες ποσότητες απορριμμάτων. Ευχαριστώ η κυρία Χάουταλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Επίτροπε που είστε εδώ σήμερα και που μας ε, κάνατε μία τόσο περιεκτική επισκόπηση των όσων κάνετε για να βοηθήσετε στο πλαίσιο των ανθρωπιστικών κρίσεων. Το πρώτο ερώτημά μου έχει να κάνει με το θέμα που έθεσε η συνάδελφος για το Ελληνίνιο. Η Μέρι Ρόμπινσον, που είναι η Γενική Γραμματέας του Ειδικού Απεσταλμένου για την Κλιματική Αλλαγή και το Ελληνίνιο, τη συνάντησα προσφάτω. και νομίζω ότι έχει πάρει πολύ σοβαρά ε, την κατάσταση και πολύ σοβαρά μας έχει προειδοποιήσει για τι καταστροφέ που θα δούμε λόγω του Ελληνίνιο και τη κλιματική αλλαγή ε, και αναρωτιέμαι κατά πόσο η Γενική Διεύθυνση Διεύθυνση ΕΚΟ έχει κάποιο πρόγραμμα για την εντόπιση των συνεπειών ε, μιας καταστροφής λόγω του Ελληνίου που θα πλήξει τις πιο ευάλωτες ε, κοινότητες. Το δεύτερο ερώτημα μου, κάπως πιο δρυμή, εντάξει βέβαια και το Ελληνίο είναι πολύ σημαντικό για το Μαλάουι, για τη Μοσούλη αναφέρατε το Ιράκ και τη Μοσούλη. Είπατε ότι η κατάσταση είναι κατά κάποιο τρόπο υποέλεγχο Υποθέτω ότι αναφέρεστε στην ανθρωπιστική κατάσταση. Όμως υπάρχουν κάποια πολύ ανησυχητικά νέα, ίσως ε, φήμες και δεύτερο χέρι πληροφόρηση ε, βιοπραγιών από το ISIS, ε, το οποίο προσπαθεί τώρα να διατηρήσει τον έλεγχο της πόλης. Τι είδους πληροφορίες έχουμε σε σχέση με αυτό. Υπάρχει κάτι που να μπορούμε να κάνουμε γιατί ακούγονται τρομερά πράγματα, αγόρια που τα παίρνουν από τις οικογένειες ε, σαν στη Σρεμπρένιτσα κάτι αλλά δέκα φορές χειρότερα. Μιλάμε λοιπόν για μια πολύ κακή κατάσταση. Τι γνωρίζουμε ακριβώς ε, ως γεγονότα δηλαδή. Μπορούμε να κάνουμε τίποτε για να παρεμποδίσουμε τέτοιου είδους ε, βιοπραγίες Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δίνω το λόγο τώρα στον Επίτροπο για να απαντήσει. Έχετε 10 λεπτά. Θα προσπαθήσω να είμαι λιτός για να μπορέσω να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις. Να ξεκινήσω από τις ερωτήσεις και τα καλά λόγια του φίλου μου Ενρίκε. Ε, θέλω να τονίσω την βασική μου πολιτική θέση ότι ως DG ECHO, ως Humanitarian Aid στην Ευρώπη θα διατηρήσουμε under any circumstances το global perspective. Γι' αυτό θα συνεχίσουμε να μιλάμε για τις forgotten crises και θα βρούμε τρόπο παρόλη την πίεση των οικονομικών να στείλουμε βοήθεια τώρα emergency στην IT και δεν θα ξεχάσουμε ούτε την Κεντρική Αμερική ούτε άλλες περιοχές του κόσμου. Ξάλλου αυτός είναι ο ρόλος μας. Να είμαστε global humanitarian actor και θα συνεχίσουμε. Θέσατε δύο-τρία ερωτήματα που αφορούν την δυνατότητα του ε, response capacity, του predictability, και του transparency. Είναι θέματα που μας απασχολούν και μέσα στην ΕΚΟ, τα συζητάμε και σε υπηρεσιακό επίπεδο πώς θα μπορέσουμε να αυξήσουμε τη δυνατότητά μας να ανταποκριθούμε. Ε, έχεις απόλυτο δίκαιο ότι το predictability είναι πάρα πολύ σημαντικό στον τρόπο που διαχειριζόμαστε την ανθρωπιστική βοήθεια. Δεν είναι πάντα τόσο εύκολο αλλά φαίνεται ότι βρίσκουμε συνεχώς ε, νέες δυνατότητες για να φτάσουμε σε ένα καλό αποτέλεσμα. Πριν λίγες μέρες ήμουν στο Πανεπιστήμιο του Λάιτεν, εδώ στην Ολλανδία, όπου έχουν ένα πολύ καλό department που ασχολείται με development και humanitarian και είδα ότι έχουν μπει κάποια πράγματα σε πιο επιστημονική βάση. Και θα βρούμε τρόπο να συνεργαστούμε και με πανεπιστήμια έτσι ώστε να βοηθηθούμε σε αυτόν τον δύσκολο τομέα. Πεατρής, ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Όπως είπα και στον Ερή και θα συνεχίσουμε και στην Κεντρική Αμερική τη βοήθειά μας. Για την Βενεζουέλα παρακολουθούμε την κατάσταση. Υπάρχουν πολιτικές ευαισθησίες, όπως καταλαβαίνετε, και η Φεντερίκα Μογκερίνη αλλά και το EAS είναι υπό συνεχή διαβούλευση και προσπαθούμε όταν χρειαστεί και προκύψει άμεση βοήθεια θα είμαστε παρόντες. Δεν υπάρχει περίπτωση να απουσιάσουμε από ενδεχόμενη ανθρωπιστική κρίση μέσα στη Βενεζουέλα. Αλλά χρειάζεται πολιτικός χειρισμός σε ό,τι αφορά τις εμπειρίες σου από την Ελλάδα. Όπως ήδη έχω πει, τα company minors είναι μία από τις τέσσερις προτεραιότητες. Ήδη οφείλω να ενημερώσω ότι η περασμένη εβδομάδα στην Αθήνα με το Save the Children είχαμε τα εγγένεια ενός πρώτου project που ασχολείται με τα ασυνόδευτα ανήλικα, τα company minors, ή στην Αθήνα ένα σημαντικός αριθμό. Είμαστε σε συνεργασία με τις ελληνικές αρχές. Ήδη κάποια καινούργια project έχουν υπογραφεί και θα μπουν σε εφαρμογή τις επόμενες μέρες. Πιστεύω ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα φτάσουμε στη μεγαλύτερη πλειοψηφία να ανταποκριθούμε σε αυτή την ανάγκη. Ε, οι υπολογισμοί και των ελληνικών αρχών αλλά και των δικών μας humanitarian partners είναι ότι περίπου έχουμε 2.300 uncompany minors στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι αν δεν είναι μέχρι τέλος του χρόνου, αρχές του νέου χρόνου, θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε, αλλά οφείλω να ομολογήσω ένα πρόβλημα. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι teenagers, είναι στην εφηβική ηλικία και είναι η πιο δύσκολη ηλικία για να τους θέσεις υπό την προστασία σου και να ελέγξεις μερικά πράγματα. Έχεις δίκιο ότι είναι η πιο τραγική πτυχή αυτής της δύσκολης κατάστασης. Προσωπικά το θεωρώ ως υπέρτατο καθήκον να δώσω ιδιαίτερη σημασία στα company minors. Και θα συνεχίσουμε. Παροτρύνουμε τους partners μας για να μας φέρουν όσα περισσότερα project να χρηματοδοτήσουμε ειδικά για αυτό το θέμα. Στα reception centers, ειδικά στα, στα νησιά, στα Aegean Islands, βρισκόμαστε σε συνεργασία με τις ελληνικές αρχές. Την κυριότερη ευθύνη βέβαια την έχει η home και ο συνάδελφος Δημήτρης Αβραμόπουλος. Ξέρω ότι ήδη αυξάνονται οι απορροφήσεις ευρωπαϊκών ε, funds για να μπορέσουν να ανταποκριθούν. Υπάρχουν δυσκολίες και στο relocation και στο resettlement. Η κατάσταση έχει εξάρσεις και οι είναι γεγονός, αλλά πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι έχει βελτιωθεί. Χρειάζεται όμως πολλή δουλειά. My dear friend έχει θέσει ένα πολιτικό ερώτημα πώς μπορούμε ως humanitarian actors ή να βοηθήσουμε ή να προλάβουμε μέσα από τις κρίσεις ή τις οικονομικές ανισότητες να προλάβουμε ανθρώπους που έχουν ανάγκη ανθρωπιστική βοήθεια. Είναι πολιτικό το ζήτημα, είναι πάρα πολύ δύσκολο πολλές φορές για τους humanitarian actors να δράσουν προληπτικά. Ε, όμως πολλές φορές η ανθρωπιστική βοήθεια εμέσως directly μπορεί να προσφέρει ακόμα και σε αυτό τον τομέα. Σεισμός στην Ιταλία. Είναι γεγονός ότι η Ιταλική κυβέρνηση δεν ε, ζήτησε την ενεργοποίηση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας, του ευρωπαϊκού μηχανισμού. Είναι επίσης γνωστό ότι η Ιταλία έχει ένα εξαιρετικό μηχανισμό πολιτικής προστασίας, ε, ίσως από τους πιο έμπειρους στην Ευρώπη, ειδικά στην αντιμετώπιση σεισμών. Βοηθήσαμε μετά από συνεργασία με τις Ιταλικές Αρχές, παρέχοντας μέσω του συστήματος Κοπέρνικους σημαντικούς χάρτες. Ε, Έχω δώσει, δώσει πολλές συνεντεύξεις σε Ιταλικά μέσα μαζιμέρωσης ενημερώνοντας γύρω από τη European Solidarity. Είμαστε σε συνεχή επαφή με τις Ιταλικές αρχές εάν χρειαστεί οτιδήποτε να δράσουμε αμέσως. Αυτό που ξέρω είναι ότι υπάρχει μια προσπάθεια τώρα να βρεθούν λεφτά από άλλα ευρωπαϊκά ταμεία ε, έτσι ώστε να δούμε αν μπορούμε να βοηθούμε στην ανοικοδόμηση ε, περιοχών οι οποίες είχαν μάλιστα ειδικό πολιτιστικό χρώμα. Ε, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν μπορώ να πω περισσότερα, δεν είναι δική μου αρμοδιότητα, αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να βρεθεί τρόπο να βοηθηθεί η Ιταλία σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Έστω και μέσω άλλων διαφορετικών ευρωπαϊκών ταμείων. Ελνίνιο. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια και ίσως χρειαστεί να κουβεντιάσουμε πριν αναχωρήσω για το Μαλάουι για να μου δώσει συγκεκριμένες πληροφορίες. Ε, έχεις απόλυτο δίκαιο όπως έχεις διατυπώσει τη θέση ότι στην περίπτωση του Ελνίνιο και του Climate Change δυστυχώς πολλές φορές κυνηγούμε την ουρά μας. Είναι μια πολύ σωστή διατύπωση ε, ελπίζω μετά το Paris Agreement να επιταχύνουμε ως ανθρωπότητα το prevention για το Ελνίνιο για να προλάβουμε νέες καταστροφές. Σε ό,τι αφορά το resilience, ειδικά στο θέμα της γεωργίας, όταν επισκέφτηκα τον Νίγηρα, είδα on the ground μια πολύ σημαντική προσπάθεια through resilience στο agriculture sector. Νομίζω μπορούμε να μεταφέρουμε αυτή την εμπειρία και σε περιοχές όπως το Μαλάουι. Ήταν όντως ε, κάτι που δεν περίμενα ότι θα είχαμε τόσο σημαντικά αποτελέσματα σε μια περιοχή, στο Σαχέλ, ειδικά στον Νίγηρα, μια από τις φτωχότερες χώρες του κόσμου. Αγαπητέ dear colleague Noiser, παρόλο που αυξήθηκαν 35% τα κονδύλια, την ανθρωπιστική βοήθεια, όπως ξέρεις και εσύ καλύτερα από μένα, ίσως είσαι πιο έμπειρος από μένα, στο humanitarian field πάλι δεν φτάνουν. Και έχω την εντύπωση ότι ποτέ δεν πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι ότι θα φτάσει η ανθρωπιστική βοήθεια στο βαθμό που θα μας ικανοποιεί ως humanitarian actors. Δυστυχώς νέες κρίσεις, νέα προβλήματα αυξάνουν καθημερινά τις ανάγκες για ανθρωπιστική βοήθεια. Είναι γι' αυτό που τονίζουμε ότι πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση και σωστά κάνει να έχει αυτό που ονομάσαμε comprehensive approach για να βρίσκει political solutions στα πολιτικά προβλήματα για να περιορίζονται οι ανθρωπιστικές ανάγκες. Δεν εκκρεμούν πληρωμές στους δικούς μας partners. Είμαστε σε πολύ καλό σημείο σε ό,τι αφορά τις πληρωμές και τις απαιτήσει. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Αυτές είναι οι πληροφορίες από όλα τα επίπεδα της ΕΚΟ αλλά είναι καλά να σας αναφέρω κάτι που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε για να ξέρετε ποια είναι τα καθημερινά προβλήματα που αναφύονται. Έχει γίνει μια μεγάλη προσπάθεια από το UNHCR στο Αφγανιστάν με στόχο το, το, repatriation process αντιλαμβάνεστε ότι σε αυτή την περίπτωση αυξάνονται αυτόματα οι ανάγκε, οι απαιτήσει. Έτσι ώστε αυτοί οι άνθρωποι όταν επιστρέψουν να έχουν τη δυνατότητα να μείνουν με δυνατότητα επιβίωση στι παλιέ του, στα παλιά τους, στα προηγούμενα, στα χωριά τους και στις παλιές τους εστίες Εδώ είναι μια αυτόματη, εντελώς ε, μη αναμενόμενη αύξηση αναγκών που προσπαθούμε να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε σε συνεργασία και in DG ECHO και in DG DEFCO για να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα. Σας είπα ένα παράδειγμα για να δώσω το πώς αναφύονται οι ανάγκες πολλές φορές εξαιτίας ειδικών συνθήκων και εξαιτίας πολιτικών συγκυριών. My dear friend, Aula, eh, thank you so much for your kind words. Σας ευχαριστώ πολύ για τα ευγενικά σας λόγια. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Και σε σχέση που είπατε με την ε, εμπειρία σας στο ελληνικό, συμφωνώ. Ότι το ελληνικό είναι ένα φαινόμενο που ε, αναμφισβήτητα δημιουργεί τρομακτικά προβλήματα και το καλύτερο το οποίο είναι και η μόνιμη μας εποδός, το μόνιμο σλόγγαν «Prevention is better than cure». Αλλά σε περιοχές οι οποίες δεν υπάρχουν υποδομές, δεν υπάρχει governance, είναι πάρα πολύ δύσκολο να χτίσεις resilience στο βαθμό που να αντιμετωπίσεις το μεγάλο impact, τη μεγάλη επίδραση του Ελνίνιο και του climate change. Μουσούλη. Επισκέφθηκα το Ερπίλ και τη Βαγδάτη τέλη Ιουλίου και έφτασα επίσκεψη πολύ κοντά στη Μοσούλη σε δύσκολες συνθήκες ομολογουμένως είδα ότι οι δικοί μας partners είχαν αρχίζει μια πολύ εντατική προετοιμασία για να προλάβουν όντως την ανθρωπιστική κρίση. Ε, μάλιστα εδώ θέλω να δώσω τα εύσημα στην κυρία Λίζ Κράντε που ήταν η συντονίστρια στην περιοχή έκανε εξαιρετική δουλειά με ένα πολύ ιδιαίτερα έντονο συντονιστικό ρόλο με όλους τους partners και όπως ξέρετε ως Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήσαμε τη βοήθεια ειδικά για το preparation, για το operation της Μοσούλης κατά 134 εκατομμύρια τον Ιούλιο και υποδέχτηκαν με πολύ θετικό τρόπο όλοι οι humanitarian actors διότι χρειάζοντουσαν αυτά τα λεφτά για το σωστό preparation. Μέχρι τώρα δεν είμαι σίγουρος ότι δεν έχω πληροφορίες ότι εμφανίζονται ιδιαίτερα προβλήματα από τους ανθρώπους που φεύγουν από τη Μοσούλη. Αντιμετωπίζεται η κατάσταση. Έχουν γίνει πολύ ε, καλά προετοιμασμένα camps, shelters, έτσι ώστε να, να μπορέσουμε να τους υποδεχτούμε. Το πρόβλημα όπως το εντοπίσατε είναι μέσα στη Μοσούλη. Και ο τρόπος που το ISIS αντιδρά στην προσπάθεια απελευθέρωσης της Μοσούλης. Οι πληροφορίες είναι όντως τόσο ανατριχιαστικές όπως τις χαρακτηρίσατε. Δυστυχώς χρησιμοποιούνται ακόμη και νέοι άνθρωποι έτσι ώστε να αποφευθεί η διείσδυση των Ιρακινών δυνάμεων μέσα στη Μοσούλη. Ξέρετε ότι είναι δύσκολο για τους humanitarian actors να δράσουν κάτω από τέτοιες συνθήκε, είναι αδύνατο. Αλλά αυτό που θέλω να βεβαιώσω, επειδή είμαι σε συνεχή επαφή και με την ε, Λίζε Κράντε, αλλά και με άλλους partners, βέβαια και με κουρδικές αρχές, μετά την επίσκεψη μου στη Μουσούλη, έχουμε αναπτύξει ένα διάλογο, αλλά και με την ίδια την Ιρακινή κυβέρνηση, τουλάχιστον στην στρατιωτική προσπάθεια υπάρχει δυνατότητα για evacuation από κάποιους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στη μέση των πυρών μεταξύ των αντιμαχόμενων παρατάξεων. Δεν θέλω να υποσχεθώ οτιδήποτε, αλλά είναι συνεχής η επαφή μαζί μας ακριβώς για να περιορίσουμε το κακό. Διότι σε τέτοιες περιπτώσεις αντιλαμβάνεστε ο βασικός στόχος είναι να περιοριστεί το κακό. Κάτι ναι, I think. Ναι. Just one minute. Ε, θέλω να δώσω έμφαση στο θέμα του global perspective που ε, ανακοινήθηκε από δύο συναδέλφους. Ε, είναι όντως σημαντικό να δώσουμε βοήθεια σε περιπτώσεις όπου ε, χρειάζεται η ανθρωπιστική βοήθεια ειδικά στο emergency phase αλλά πρέπει να κάνουμε ένα διαχωρισμό μεταξύ του humanitarian και του development. Αλλιώς εάν δεν καταφέρουμε να το διαχωρίσουμε δεν θα μπορούσαμε και να συνεργαστούμε αποτελεσματικά. Οι humanitarian actors με τους development actors. Και μια τέτοια περίπτωση είναι η IT. Σίγουρα θα προσπαθήσουμε μέσα στον περιορισμό, μένω την περιορισμένη δυνατότητα την οικονομική να δώσουμε βοήθεια τώρα στην ΑΕΤ, αλλά σίγουρα μαζί με την ΤΕΦΚΟ θα είμαστε σε συνεννόηση έτσι ώστε να συνεχίσει ως development activities or development aid. Θέλω να κλείσω με ένα υπενιγμό που άφησα στην αρχή ότι το European Project βρίσκεται για πρώτη φορά σε τόσο critical juncture, σε τόσο σημαντικό σταυροδρόμιο challenge. Την ίδια στιγμή όμως, επειδή εκτός από την Αφρική και άλλες περιοχές κάνω και μια περιοδία για να συναντήσω τις αντίστοιχες κοινοβουλευτικές επιτροπές μέσα στην Ευρώπη, ήμουν στην Ιρλανδία τελευταία και αλλού, βλέπω ένα σημαντικό τμήμα της ευρωπαϊκής κοινή Νόμης και των ευρωπαίων πολιτικών σε κάθε member state να δείχνει μια διάθεση και αποφασιστικότητα ότι παρόλα τα προβλήματα, παρόλες τις ελλείψεις, το European project remains the only way for the whole Europe Το ευρωπαϊκό εγχείρημα αποτελεί το μοναδικό δρόμο για την Ευρώπη και για όλους εμάς ως Ευρωπαίους. Ευχαριστώ πολύ. Thank you, Colleagues, item 20. Ευχαριστώ. Για το 21 δεν υπάρχουν ερωτήσεις, για το 22 δεν υπάρχουν διάφορα. 23 επόμενη συνεδρίαση 28 Νοεμβρίου επόμενη πλήρη συνεδρίαση και 29 Νοεμβρίου. Υπάρχουν κάποιες επιπλέον συνεδριάσεις και εργαστήρια. Θα σας αποστείλουμε ένα σημείωμα. Ενδεχομένω μπορεί να υπάρξει και τετάρτη απόγευμα συνεδρίαση στο Στρασβούργο με την Φεντερίκα Μογκερίνη. Θα σας ενημερώσουμε. Θα σας ενημερώσει η Γραμματεία για όλες τις επιπλέον ε, συναντήσεις. Ε, πολύ ενδιαφέροντα και αυτά που συμβαίνουν εκατέρωθεν του Ατλαντικού. Φαντάζομαι ότι θα τα παρακολουθήσετε κι εσείς. Ε, ευχαριστούμε και τους διερμηνείς και ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον Επίτροπο για την παρουσία του σήμερα.